Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Καθίστε σας παρακαλώ και εσείς κύριε Λιγκρυπ. Να ξεκινήσουμε. Πρέπει να σας ε, πω ότι ε, πρώτα απ' όλα ε, έχουμε την συνεδρίασή μας η οποία θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Επίσης μου είπαν οι μυστικέ μου υπηρεσίε ότι είχε γενέθλια χθε ο αντιπρόεδρο Μαρτίνες. Γι' αυτό λοιπόν του ευχόμαστε τα καλύτερα και στην προσωπική του ζωή και εδώ στην Επιτροπή μας. Έχετε ήδη από την 19η Ιανουαρίου την ε, ημερήσια διάταξη. Όμως το πρόγραμμά μας έχει υποστεί τρομερές αλλαγές. Πρώτον, διότι η κυρία Γιαννάκου e είναι άρρωστη και δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας ούτε σήμερα ούτε αύριο. Είναι δε η συγκήτρια για το θέμα των, των πολιτικών κομμάτων και, και τη χρηματοδότησή τους. Και επομένως θα πρέπει να αφαιρέσουμε το σημείο αυτό από τη μέση διάταξη. Επίσης, μετά από τη σημερινή μα συνεδρίαση, θεωρητικώς, θα έπρεπε να έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Δυστυχώς όμως κάποιοι ε, από τους συντονιστέ δεν μπορούν να είναι παρόντες σήμερα, οπότε θα την κάνουμε αύριο το πρωί. Η συνεδρίαση λοιπόν των συντονιστών θα γίνει αύριο το πρωί. Επίσης, οι συνεισηγητές ε, για την ε, πρόταση τροποποίηση των συνθήκων δεν μπορεί να είναι αύριο πριν από τις 10.30 μαζί μας. Επομένως, θα ξεκινήσουμε 9 η ώρα με τους συντονιστές και στις 10.30 θα συνεχίσουμε με το σημείο της σημερινής διάταξη που αφορά την τροποποίηση των συνθήκων. Επομένως, στην ουσία, σήμερα... Το μόνο που μας παραμένει, παραμένει στο πρόγραμμά μας είναι η εξελίξη στην ΚΟΖΑΚ, καθώς επίσης και η δικιά μου έκθεση για την ερμηνεία του άρθρου 51, ενώ ε, η, η έκθεση για την οποία είμαι εισηγητής. Αύριο λοιπόν θα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών και μετά θα έχουμε και την Αντιπρόεδρο Διάνα Γουόλης η οποία θα έχει μαζί μας μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα κοινό μητρό διαφάνειας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Mm, mm, Υπό τα διάφορα, εγώ θα ήθελα να προσθέσω και ένα θέμα το οποίο αφορά ε, την ε, ε, τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 216 του κανονισμού διότι οι τέσσερις συνεισηγητές και της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Αναφορών συμφωνούν αλλά και άλλα θεσμικά όργανα συμφωνούν. Συμφωνούν, λέγω, ότι υπήρξε λάθος στην τελική έκθεση και αυτό το τυπικό λάθος θα πρέπει να διορθωθεί. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό αύριο. Επομένως τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως ή μάλλον το δεύτερο σημείο. Στο, αναφέρομαι τώρα στην ε, τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών, 13 της Δεκεμβρίου και 12ης ε, ε, Ιανουαρίου. Εκεί αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει έκθεση Σμιτ ε, όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο νομοθέτησης. Επίσης, βάσει εφαρμογής του άρθρου 123 του κανονισμού, θα έχουμε έναν εισηγητή από το ΕΛΚ, ακόμα δεν έχει οριστεί το όνομά του. Όσον αφορά τώρα την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 128 του κανονισμού δηλαδή την, ε, ε, την προάσπιση των ε, εξαιρέσεων του και δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου ενώπιον του δικαστηρίου. Αυτό θα εξεταστεί από τον υποφαινόμενο. Ο κύριος Γκουερέρο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις ε, όσον αφορά την ε, ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ θα προσκληθεί για να παρουσιάσει σε μια επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας τα τελευταία έγγραφα όσον αφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι πρόεδρος της Επιτροπής εδώ συμμετέσχων εις την συνεδρίαση μιας διοργανικής ομάδας ε, σχετικά με την ε, θέση σε πρακτική ισχύ της κοινή δήλωσης της 9 Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Μαζί για την καλύτερη επικοινωνία στην Ευρώπη». Τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη και αυτό ε, υπόθηκε εκεί. Ε, επίσης να πούμε ότι το 2011 θα είναι ε, το ευρωπαϊκό έτος για τις ευρωπαϊκές δράσεις και το 2012 δεν θυμάμαι τι θα είναι, λέει ο Πρόεδρος, για τους ηλικιωμένους. Δεν μας αφορά αυτό φυσικά λέει ο Πρόεδρος γιατί είμαστε όλοι νεότατοι. Α, το 13, το 2013 θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, μάλιστα. Και στα πλαίσια των ε, συντονιστών θα δούμε εν λεπτομερία ποια είναι τα στοιχεία τα οποία εμείς μπορούμε να προτείνουμε έτσι ώστε στα πλαίσια αυτής της σημαντικής ε, δράσης να έχουμε και εμείς ε, τον λόγο μας και να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα και εν τέλει γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρακτικά σας έχουν ήδη μοιραστεί και βρίσκονται στη διάθεσή σας ε, και εάν ε, δεν υπάρχουν σχόλια ε, σύμφωνα με το Ιωθώτα, θα, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά των συνεδριάσεων 8 9 Νοεμβρίου του 2010, 29-30 Νοεμβρίου 2010, 13 Δεκεμβρίου 2010. Περνούμε επομένως στο σημείο 4. Εξελίξεις σχετικά με την ΚΟΖΑΚ. Όπως σας είπα και από την αρχή, έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο Μιγελ Άγχελ Μαρτίνες, ο οποίος έχει μια πρώτη συνάντηση την, 5η Οκτωβρίου. Και θα κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στην ΚΟΖΑΚ. Τι έγινε μέχρι τώρα και ποιες είναι οι προβλεπόμενες εξελίξεις για το μέλλον. μαζί με τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες ε, ε, ξέρουμε ότι ε, πέρασε και η τροποποίηση του άρθρου 139 ε, και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ε, την ρόμη του Αντιπροέδρου Μαρτίνες και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συζητά για θέματα εξαιρετικά ε, σημαντικά και ευαίσθητα. Επίσης να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση ΚΟΖΑΚ σε επίπεδο Προέδρων Επιτροπών θα λάβει χώρα την 10η και 11η Φεβρουαρίου στη Βουδαπέστη ενώ η συνεδρίαση ΚΟΖΑΚ θα γίνει 29 και 31 μέχρι 31 Ιού πάντα στην Βουδαπέστη. Σας δίνω το λόγο λοιπόν κύριε Μαρτίνες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πάντατε, βέβαια για μένα συνιστά ιδιαίτερη ικανοποίηση η πρόσκληση να παρευρεθώ στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και στην προκειμένη περίπτωση έρχομαι εδώ όχι μόνο υπό την ιδιότητά μου και την αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου και την ΚΟΣΑΚ, αλλά παρεμβαίνω και υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Διευθυντικής Επιτροπής, αν θέλει της Επιτροπής Καθοδήγησης, Steering Committee, που θα παρακολουθήσει ό,τι έχει να κάνει με την πρακτική εφαρμογή της συνθήκη της Λισαβόνας σε σχέση με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και τη συνεργασία τους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Καζίνη που μου ευχήθηκε για τα γενέθλιά μου. Και να πω και στον ίδιο και σε εσά του υπόλοιπου ότι αυτό το οποίο συγκροτήσαμε είναι μια ομάδα προβληματισμού. Στόχος του είναι να ε, μετράμε την ηλικία στα γαλλικά, επειδή τα 60 κρατάνε 10 χρόνια ε, στα γαλλικά. Τελικά καταλαβαίνει ότι η όταν ήταν φτάσει στα 80 με τα γαλλικά. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνεδρία, θα σα πω εγώ λίγο πώ πήγαν τα πράγματα με την Κόσα και στο τέλο θα με επιτρέψετε να κάνω έτσι δύο-τρία πιο προσωπικά σχόλια, πιο, να σας μεταφέρω πιο προσωπικές μου σκέψεις σε σχέση με το ότι εδραιώνουμε και τις σχέσεις μας με την Κόζακ και τη μόνιμη ομαλή και ροή σχέσεων που έχουμε και θα δούμε και σε σχέση με το μέλλον τι προβλέπει. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι πολύ που έχω στο πλευρό μου τον πρόεδρο Καζίνη και συνεργάζομαι μαζί του διότι η συμβίωσή μας είναι πάντοτε τέλεια και άλλοι υποστηριζόμαστε, αντλούμε ο ένας δύναμη από τον άλλο. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Όπως γνωρίζετε, στην τελευταία τροποποίηση του κανονισμού θεσπίστηκε ότι μαζί με τον ε, κύριο Καζίνη θα προεδρεύουμε της αντιπροσωπείας που στέλνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ε, συνεδριάσεις της ΚΟΖΑΚ. Στην τελευταία συγκεκριμένα συνεδρίαση είχαμε μαζί μας και τέσσερις συναδέλφους οι οποίοι θα εμπλούτιζαν ιδιαίτερα τις εργασίες εκεί. Μακμίλαν Σκοτ, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Περβόν Μπερές, Μέσερ Σμιτ, που είναι και εδώ και διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή του, και Έλμαρ Μπροκ. Αυτοί ήταν οι τέσσερις συνάδελφοι. Εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς ε, αιτιολόγησε την παρουσία του με τα θέματα τα οποία προβλέπονταν στην ημερησία διάταξη των συζητήσεων, οικονομική διακυβέρνηση, κοινή πολιτική επίσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ποιε είναι οι εντυπώσει που έχω συναγάγει εγώ ή μου λέει η γραμματεία γραμματεια έχω συναγάγει. Στη συνεδρίαση που έγινε στις Βρυξέλλες υπήρξαν καρποφόρες ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων για θέματα πολύ σημαντικά όπως είναι η οικονομική διακυβέρνηση, η στρατηγική 2020, η αηφόρος ανάπτυξη. Και νομίζω ότι ενδιαφέρουσες ήταν και ανταλλαγές απόψεων στην ε, επιτροπή, στις επιτροπές ε, με τον Λετέρ, με τον Μπαρόσο και με τον Φον Ρομπάι. Μου δίνεται η εντύπωση ότι στην Κόζακ υπάρχει μια τάση να μην μείνουν στα θέματα τα ε, θεσμικά, επικαιρικότητας, ε, επικουρικότητας ή κάποια άλλα θέματα πιο οργανωτικά και η ΚΟΖΑΚ να ασχοληθεί περισσότερο με μεγάλα οριζόντια θέματα όπως είναι η κατάσταση της Ένωσης ή το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε γενικές γραμμές, τα κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν σε αυτή την ε, συνεδρίαση το κείμενο συγκεκριμένα που λέγεται ε, η συμβολή και το άλλο το κείμενο με τα συμπεράσματα, νομίζω ότι περιέλαβαν και κάποια σχόλια και τροπολογίες από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευτυχώς λοιπόν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες και ιδίως ό,τι αφορά την διακοινοβουλευτική παρακολούθηση, τον διακοινοβουλευτικό έλεγχο σε θέματα πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ο Έλμαρ Μπρόκ εκεί έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και τελικά εγκρίθηκε και ένα κείμενο που νομίζω ότι είναι αποδεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια πάντοτε υπάρχει η κατάσταση που δεν είναι και τόσο ευχάριστη για την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, συχνά εμφανίζεται ένα αρχικό κείμενο που δεν είναι καθόλου αρεστό για την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρεστό και υπό την έννοια ότι είναι σαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ήταν ένα ξένο σώμα στην Κόζακ. Ε, και μετά, μετά από πολλές τροπολογίες και πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές έτσι, επαφές, φιλικές κτλ. Αυτό το οποίο στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το δεχθούμε, κάπως ε, τακτοποιείται. Έτσι λοιπόν, ε, ξεκινάμε πολύ άσχημα και μετά ε, είναι κάπως ε, αποδεκτό, κάπως ανεκτό, θεωρείς ότι είναι και καλό. Μα δεν είναι έτσι, γιατί τελικά εγκρίνονται κείμενα που εντάξει, εάν τα ενέκρινε κάποιος εκτός θα ήταν καλά. Αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να δεχθούμε ένα κείμενο που απλά κατά κάποιο τρόπο το θεωρούμε ανεκτό. Και είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, υπήρξε από την άλλη πλευρά ένα σημαντικός αριθμός μεγάλων εντάσεων, στιγμών μεγάλης έντασης λόγω μιας καθαρά εχθρική θετική στάσης από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια. Και κυρίως αυτό αφορούσε τη διοργανική συμφωνία. Τη διοργανική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή. Τελικά, το κείμενο που προέκυψε από όλη αυτή τη συζήτηση δεν είναι ένα κείμενο που εμείς δεν θα είχαμε μπορέσει να προσπογράψουμε. Εμένα όμως αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι η σαφώς, η καταφανώς εχθρική στάση ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων. Και συγκεκριμένα του συναδέλφου τη Φινλανδίας, και όχι μόνο του συναδέλφου από συντρόφου έτσι του θεωρώ εγώ, συντρόφου τη δική μου ιδεολογική οικογένεια. Πάρα πολύ επιθετική ήταν η στάση του. Το πρόβλημα όμω δεν είναι τόσο ότι μπορεί να υπάρχει ένα κοινοβούλιο το οποίο οι εκπρόσωποι συμπεριφέρονται εχθρικά προς το Ευρωκοινοβούλιο. Το πρόβλημα είναι ότι τον Φιλανδό να τον μιμηθεί ένα Σουηδός πάλι από τη δική μου νομίζω πολιτική οικογένεια και να έχουν την ίδια στάση, την ίδια θέση. Αυτό ξέρετε με ανησύχησε λίγο περισσότερο και γενικώ προκαλεί περισσότερη ανησυχία. Μπορεί να εκπλήσει λιγότερο, αλλά ανησυχεί περισσότερο το ότι και κάποιοι Βρετανοί εκπρόσωποι συμπαρατάχθηκαν σε αυτή την κινητοποίηση, αν θέλετε. Οπότε εκεί η έκπληξη ε, ε, είναι αρκετή και ακόμη μεγαλύτερη γίνεται όταν έχουμε και Ολλανδούς συντρόφους, αλλά όταν οι και εκπρόσωποι της Bundestag ακολουθούν την ίδια γραμμή, τότε τρελαίνεσαι. Αυτό επίσης που εκπλήσει είναι ότι ίσως λόγω σε πνεύμα έτσι καλής ε, ανατροφής, επίδειξης καλής ανατροφής και καλής παιδείας, οι υπόλοιποι σιωπούν, μένουν άλλαλοι. Ή σιωπούν ή τόσο πολύ ελάχιστα δείχνουν να διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτά που λέγονται, που τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μένει μόνο και απομονωμένο. Σαν να επρόκειτο για εχθρούς, για αντιπάλους. Ενώ, όπω είπα στην αρχή, υποτίθεται ότι στην Κόζακ όλοι πηγαίνουμε προ την ίδια κατεύθυνση και ότι όλοι αυτό που επιδιώκουμε είναι η συμπληρωματικότητα και οι καλέ σχέσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά στο τέλος θα σας κάνω και κάποια σχόλια έτσι εμβαθύνοντας περισσότερο. Τώρα, νομίζω ότι υπήρξαν και κάποια σημαντικά στοιχεία, πολύ σημαντικά. Όπως σας είπα, φτάσαμε σε μια αποδεκτή συμφωνία σε ό,τι αφορά το διακοινοβουλευτικό έλεγχο και παρακολούθηση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και κατά πάσα περίπτωση στην διάσκεψη των Προέδρων που θα λάβει η χώρα σε αρχές Απριλίου, εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει σημαντική πρόοδος, ξεκάθαρη πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Οι φίλοι Βέλγοι έχουν αναλάβει νομίζω την επεξεργασία αυτού του θέματος και πραγματικά τρέφω πολύ μεγάλες ελπίδες για το ότι θα έχουμε μια πολύ ή έστω αρκή, αρκετά ικανοποιητική για εμάς εξέλιξη και συνεργασία. Υπάρχουν σημαντικά θέματα που δεν είναι επίμαχα, θα έχουν συμπεριληφθεί και στι επόμενε διακοινοβουλευτικέ συναντήσει αυτά τα θέματα, στη, ό,τι αφορά την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, η Europol, Eurojust, την ασφάλεια και το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλω να σας πω και να αποτίσω και φόρο τιμής ταυτόχρονα στο ρόλο των δύο βουλών άνω και κάτω βουλής του Βελγίου. Διότι το Βέλγιο πολύ αποφασιστικά αντιμετώπισε και αντιστάθηκε στις άλλες παρεμβάσεις πάρα πολύ αποφασιστικά σε σημείο που σε κάποιες περιπτώσεις ανετράπησαν αποτελέσματα ψηφοφοριών και έτσι ε, κάποια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί ε, χάρη στους Βέλγους που βάλαν, θέλετε, όλο το κάρβουνο και στην ατμομηχανή. Άλλα κοινοβούλια, Ιταλοί, να δώσω ένα παράδειγμα, κάποιοι Γάλλοι συνάδελφοι, κάπως ακολούθησαν αυτή την πιο λογική γραμμή θα έλεγα, για να μην χρησιμοποιήσω πολιτικούς όρους. Απλά να πω ότι κάπως έτσι ε, πιο σωστή διόρθωση της συμπεριφοράς και της τάσης σχέση με άλλους συναδέλφους τώρα. Τώρα, τι θα γίνει επί Ουγγρικής Προεδρίας. Ο πρόεδρος Καζίνη και εγώ προσωπικά πριν από τρεις ή τέσσερις ημέρες νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα Είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, της Ουγγρικής Βουλής και με τον ε, αρμόδιο εξωτερικών υποθέσεων και ο υπεύθυνο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις θα προεδρεύσει και τις συνεδρίασεις της ΚΟΖΑΚ στη Βουδαπέστη η συνάντηση επίσης των, και στη συνάντηση των Προέδρων και στην Ολομέλεια το Μάιο, 1931. Νομίζω ότι ήταν επικοδομητική, θετική και εγκάρδια η συνάντηση που είχαμε με τους ε, συναδέλφους μας. Είπαμε ότι πρέπει να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, με την Ουγγρική Προεδρία και ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μας έδωσε ένα αίτημα του Δανικού Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου της Δανίας, που έλεγε ότι στις συζητήσεις της ΚΟΖΑ καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί ο όρος της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας. Ήταν ένα αίτημα αυτό από πλευρά Δανία. Για να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση που κάποιοι άλλοι είχαν προτείνει, δηλαδή να θέσουμε την Ουγγρική Προεδρία ε, ενώπιον τη δύσκολη βέβαια ε, θέση να προβεί σε αυτοκριτική. Από ό,τι κατάλαβα και από πλευράς, μάλλον νομίζω και από πλευράς Καζίνη, ε, η απάντηση που δώσαμε είναι ότι είμαστε σύμφωνοι με την Ουγγρική πλευρά ότι δεν εμπίπτει το σημείο αυτό και το αίτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη, η οποία είχε προκαταρτιστεί. Δεν θέλουμε να υπάρξει σύγκρουση και αντιπαράθεση, αλλά να επιτευχθεί πρόοδος. Και βέβαια, σε κάποια χρονική στιγμή όλοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους με τον τρόπο που θεωρούν πιο σωστό. Μια άλλη επιστολή πάλι από το Κοινοβούλιο της Δανίας για μια ακόμη φορά έκανε λόγο στο θέμα των γλωσσών, της πολυγλωσσίας που είναι πολύ σημαντικό και για μένα και με αφορά γιατί είμαι και ο αρμόδιος αντιπρόεδρος για θέματα πολυγλωσσίας. Και το Δανικό Κοινοβούλιο πρότεινε να εργαζόμαστε στα αγγλικά και τα γαλλικά και γιατί θα εξοικονομούσαμε χρήματα κτλ. κτλ. Και φυσικά αυτό είναι ριζικά αντίθετο στην πρακτική ως θέμα αρχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποια στιγμή βέβαια είπα, το είπα και εγώ, ότι εμένα δεν θα με ανησυχούσε ε, να μιλάμε σε δύο μόνο γλώσσες, αρκεί κανένας να μην μιλάει τη μητρική του γλώσσα, για να είμαστε όλοι επίσης όρις. Ωραία, να μιλάω εγώ αγγλικά ή γαλλικά, αλλά οι Γάλλοι να μην μιλάνε γαλλικά και οι Άγγλοι να μην μιλάνε αγγλικά. Για να μην μιλάμε ε, κάποιοι τη μητρική μας γλώσσα και κάποιοι άλλοι όχι. Δεν είναι καλό να περιθωριοποιούνται ε, γλώσσες, να περιθωριοποιείται η χρήση γλωσσών και να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα κάποιες άλλες χώρες πέραν του ότι η χρήση της γλώσσας είναι και στοιχείο της ταυτότητας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα δοκιμήσει αυτή η πρόταση. Ο πρόεδρος τώρα Κασίνη πρότεινε και με είχε τις, πλήρου ε, ε, τις πλήρους υποστήριξη πρότασή του να συζητηθεί το θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών, της πρωτοβουλίας των πολιτών καθώς και το θέμα του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Νόμου. Όμως η Τρόικα της τελευταίας Κόζακ προς το παρόν φαίνεται η φάνη και τέλος πάντων να μην είναι ευνοϊκά διακείμενη απέναντι σε αυτές τις προτάσεις. Εγώ νομίζω, αν συμφωνεί και ο κύριος Καζίνη, ότι μπορούμε να επανυποβάλουμε τα αιτήματα αυτά. Ο πρόεδρος Καζίνη επίση είπε ότι πρέπει να δούμε και το θέμα της θρησκευτική ελευθερίας. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα, θα μιλήσουμε για την κατάσταση της Ένωσης, ε, παρουσία του Πρωθυπουργού Όρμπαν, του Πρωθυπουργού Μπαρόσο και του Αντιπρόεδρου Σεύκοβιτς. Θα μιλήσουμε για τη στρατηγική 2020, οικονομική διακυβέρνηση, ευρωπαϊκό εξάμεινο, πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2012 και θα ακούσουμε επίσης την έκθεση της Βελγικής Προεδρίας σε σχέση με τη διάσκεψη των Προέδρων των αρχών Απριλίου. Τώρα, εν κατακλείδη, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που αντιλαμβανόμαστε στις σχέσεις μας με την ΚΟΖΑΚ. Αλλά οι δυσκολίες αυτές ουσιαστικά είναι, σχέσεις, ε, είναι μάλλον δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις σχέσεις μας με τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν έχει να κάνει με την ταυτότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυσκολία αυτή, αλλά με την ταυτότητα των εθνικών κοινοβουλίων οι συντάκτες, που είμαστε εμείς ίδιοι δηλαδή, πιστεύαμε ότι θα είχαμε να συναντήσουμε 27 εθνικά κοινοβούλια. Τελικά συναντηθήκαμε με 40 βουλές. Υπάρχουν ε, μια σειρά χωρών που είπαν ότι έχουν περιφερειακά κοινοβούλια που έχουν αποκλειστική νομοθετική αρμοδιότητα. Εγώ νόμιζα ότι αυτό ίσχυε μόνο για τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Αλλά απατηθήκαμε. Είδαμε ότι και στην Πορτογαλία υπάρχουν περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές αρμοδιότητες. Το ίδιο ισχύει στη Φινλανδία, με το Έλαντ, το νησί Έλαντ. Και άρα τελικά ο αριθμός 40 μπορεί να γίνει και 120. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι ε, πνίγουμε το ψάρι στο νερό που λέει ναι, και οι Γάλλοι φίλοι μου. Δηλαδή κάνουμε τα πράγματα πάρα πολύ πολύ πλοκά. Έχουμε τις νήσους Φερόε από τη Δανία, μπορούμε να έχουμε και κοινοβούλια και στο Ενωμένο Βασίλειο που θα προκύψουν. Ε, το σκοτικό κοινοβούλιο, τέλος πάντων, περιπλέκεται πάρα πολύ κατάσταση. Περιπλέκεται και για την, λόγω της ε, ανομοιογένεια των εθνικών κοινοβουλίων και σε ό,τι αφορά το μεγεθό τους και σε ό,τι αφορά το πόσο ενδιαφέρονται ή όχι για τα ευρωπαϊκά θέματα και τη δυνατότητα που έχουν να κάνουν αυτά που λέει η συνθήκη της Λισαβόνας, ε, ίσως έχουν, υπάρξουν κάποιες αρμοδιότητες, κάποιες ευθύνες, Υπάρχει και ένα πρόβλημα που δεν είναι βέβαια των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά ένα είδος ευρωσκεπτικισμού, που πάντω κάπως προβάλλεται και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Πάντω, νομίζω ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος φέτος, ιδίως ό,τι αφορά τον εξορθολογισμό των σχέσεων. και υπήρξε και πολύ σημαντική συμβολή και των μελών της Επιτροπής σας. Νομίζω ότι καταφέραμε κάπως να συντονίσουμε Δηλαδή όχι να έχουμε πέντε συναντήσεις ένα μήνα και τους επόμενους δύο να μην έχουμε καμία. Εγκρίναμε λοιπόν και το πρόγραμμά μας, ε, το πρόγραμμα της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας του Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα χρόνο και σε σχέση και με την Κομισιόν και νομίζω ότι ήταν ικανοποιητική και λογική η πρόοδος που σημειώσαμε στον τομέα αυτό. Ολοκληρώνοντας θα μου επιτρέψετε να σας σχολιάσω το πρόβλημα ουσίας το οποίο αντιμετωπίσαμε. Και θα ήθελα να αφιερώσω και ένα λεπτό στις ε, εναλλακτικέ που βλέπω εγώ για το μέλλον. Λοιπόν, το πρόβλημα το οποίο τίθεται προέρχεται από το όραμα, αν θέλετε, κάποιων ε, κρατών που υπάρχει, εγώ δεν το βλέπω σωστό, που λένε ότι όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατακτά μεγαλύτερες ποσοστώσεις αρμοδιοτήτων, εξουσιών, αυτό συνιστά ένα βήμα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αυτό μου φαίνεται λάθος γιατί εγώ πάντοτε νόμιζα και πίστευα ότι ο εκδημοκρατισμός της διαδικασίας ευρωπαϊκής οικοδόμησης μετράται κατά κύριο λόγο με την ε, αύξηση, τη συνεχή αύξηση από συνθήκη σε συνθήκη των εξουσιών που κατακτά, που αποκτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και φυσικά κάθε φορά που κατακτά, αν θέλετε, ε, κάποιου είδου μεγαλύτερη εξουσία λήψη αποφάσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σίγουρα αυτό γίνεται σε βάρος του μονοπωλίου λήψη αποφάσεων που είχε το Συμβούλιο μέχρι τότε στου διάφορου τομεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό το οποίο ποτέ εγώ δεν είχα διανοηθεί είναι ότι σε κάποια εθνικά κοινοβούλια υπήρχε η σκέψη και η αντίληψη ότι αυτή η μεγαλύτερη εξουσία συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λιγότερο μονοπόλιο του Συμβουλίου θα ήταν για τα εθνικά κοινοβούλια να βγουν προς τα πίσω, διότι θεωρούν ότι αυτά, τα εθνικά κοινοβούλια δηλαδή, ελέγχουν το Συμβούλιο μέσω του ελέγχου, υποτίθεται ότι ασκούν επί των εκάστοτε και των κυβερνήσεών τους που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο. Ήμουν 22 χρόνια εθνικός βουλευτής. Ήμουν και εκπρόσωπο σε θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων. Και εξωτερικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούστε, ήμουν και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση εκπρόσωπος και ξέρω ποιο είναι το επίπεδο ελέγχου που οποιοδήποτε Εθνικό Κοινοβούλιο ασκεί πραγματικά επί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εξού και πραγματικά φαίνεται εντελώ παράλογο, εκτός λογικής να σκέφτεται κανείς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες αυτό συνεπάγεται ότι χάνεται ο δημοκρατικός χαρακτήρας ε, της όλης διαδικασίας. και έχουμε αυτούς ε, που ε, εκφράζουν κάποιες αντιρρήσεις και αντιστέκονται για αυτό το λόγο και σε αυτούς έρχονται να προσθεθούν οι ευρωσκεπτικιστές και όλοι όσοι αντιστέκονται σε όλα. Και το βλέπουμε και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια και παντού βλέπουμε κάποιους να έχουν και να επισύουν την κάρτα που λέει όχι για όλα, για τα πάντα. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε και νομίζω ότι θα πρέπει, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αλλά με ιδιαίτερη προσοχή και λεπτότητα αυτό το ζήτημα. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι υπάρχουν δύο προβλήματα που τίθενται και για τα οποία πρέπει να βρούμε λύση. Το πρώτο πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που ευτυχώς το, το είδα λιγότερο στις Βρυξέλλες και είμαι σίγουρος ότι συμφωνεί και ο Καζίνη μαζί μου. Είναι το πρόβλημα που έχει να κάνει με το ότι τα εθνικά κοινοβούλια και η Κομισιόν με τους τεράστιους πόρους της ε, ε, Κομισιόν προσπαθούν να φτιάξουν μια γέφυρα ενός υποτιθέμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου, ελέγχου της Κομισιόν από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό λογικά σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακάμπτεται κατά κάποιο τρόπο και είναι και ενάντιο στη διαδικασία που θεσπίζει η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό που ήθελαν κάποια κοινοβούλια είναι να αποτελέσουν ε, ένα δεύτερο, ίσως τρίτο κοινοβούλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είχε απορριφθεί όταν είχε τεθεί κατά το παρελθόν. αυτό το πρόβλημα που ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα γιατί από πλευράς Κομισιών ήταν σαφές ότι υπήρχε η τάση να είναι αρεστή στα εθνικά κοινοβούλια και να έχει έτσι κάποιες επαφές και δεν μιλάω μόνο για τον πρόεδρο, μιλάω για οποιονδήποτε επίτροπο, επιτροπογεωργίας, που πηγαίνει στις επιτροπές, στις αρμόδιες των Εθνικών Κοινοβουλίων, ο επίτροπο, Μεταφορών που πηγαίνει στην Επιτροπή Μεταφορών των Εθνικών Κοινοβουλίων κτλ. Δηλαδή να υπάρξει ένα δίκτυο επαφών που φυσικά και απριόρι δεν μπορεί να το δει κανείς ως κάτι αρνητικό, αλλά εάν αυτός ο μηχανισμός τελικά αποσκοπήσει στην αντικατάσταση, στην υποκατάσταση της διαδικασίας που προβλέπει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον έλεγχό του απέναντι στην Κομισιόν, τότε δημιουργεί πρόβλημα. Ο πρόεδρος Μπαρός ήταν πολύ ξεκάθαρος, πολύ αποφασιστικός και πάρα πολύ φιλικός προς το Κοινοβούλιο στην συνάντηση της Κόζαξ στις Βρυξέλλες. Πραγματικά εξαιρετικά, εγώ ποτέ δεν τον είχα ακούσει να μιλάει με τόσο μεγάλη σαφήνεια απέναντι σε ένα καθαρά εχθρικό έτσι περιβάλλον. Ούτε τόσο ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που μπορώ να σας το πω αυτό. Διότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ αποφασιστική παρέμβαση. Και επαναλαμβάνω ότι δεν ήταν και τέτοιο το κλίμα που να μπορού, μπορούσε εύκολα να είναι κανείς τόσο αποφασιστικός. Το έκανε όμως ο πρόεδρος Μπαρός. Το δεύτερο πρόβλημα που θέλω να φέρω έχει να κάνει κυρίως με το πώς θα οργανώσουμε κάτι το οποίο προβλέπεται από τις συνθήκες ε, παρακολούθηση, για να μην πω έλεγχος, της εξωτερικής πολιτικής ε, και της, πολιτικής, ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Εδώ βλέπουμε επίσης ένα περίεργο φαινόμενο. Δηλαδή, αναφέρεται, γίνεται αναφορά ε, στην ε, ε, στη συνέλευση του Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά αυτή πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Εγώ ήμουν 14 χρόνια αντιπρόεδρος της συνέλευσης και 20 τόσα χρόνια μέλος. Φυσικά και δεν είπα ότι δεν ήταν μια οντότητα που είχε σημασία. Φυσικά και είχε. Αλλά να λέει κανεί σήμερα ότι η συνέλευση αυτή ασκούσε τον έλεγχο ασκούσε έλεγχο στις κυβερνήσεις και στα κράτη σε ό,τι αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι πλήρης διαστρέψης πραγματικότητας. Μιλούσα και με τον Βέλγο, με τον, τον πρώτο της Βελικής Συνέλευσης και το έλεγα, όταν εσείς ήσασταν υπουργό Άμυνα, που ήταν επί 20 χρόνια υπουργό Άμυνα, άρα του είπα, όταν εσείς πηγαίνατε στην κοινοβουλευτική συνέλευση της Ευρωπαϊκή Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, σας Έλεγξε κάποιο, κατά το ελάχιστο έστω. Όχι βέβαια μου λέει, εμεί απλά πηγαίναμε εκεί, μιλούσαμε, τα εξηγούσαμε, τα λέγαμε. Αυτό γινόταν τότε. Δεν υπήρχε έλεγχο. Το θέμα είναι λοιπόν, τι τι θα κάνουμε τώρα. Και εδώ έχουμε μια πρόκληση. Συνάδελφοι της Επιτροπής όπως ο ε, κύριος ε, Γουαλτιέρη, ο κύριος Νταφ, δεν ξέρω αν είναι ε, μέλος της Επιτροπής, αλλά είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης ούτως ή άλλως, όπως και ο κύριος Μπροκ. Πώς, τι θα προτείνουμε, τι θα πούμε. Το βελγικό... Έχουμε μια βελγική πρόταση και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως, όπως και να έχει, σε σχέση και μαζί με αυτή την πρόταση, αυτή την πρόταση της Βελγικής Προεδρίας, που θα πρέπει να εξετάσουμε και να υποβάλουμε ή να μην υποβάλουμε τροπολογίες, μαζί με αυτό λοιπόν έχουμε ένα εγγραφό το οποίο εξουσιοδοτεί ένα ε, κοινοβούλιο εθνικό που δεν θέλω να κατονομάσω για να μην γίνω αντιπαθής, του οποίου η επιθετικότητα κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φτάνει ε, στα, στα όρια, να προτείνει όταν συνεδριάζει στις Βρυξέλλες ο οργανισμός που αυτοί λένε να μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε πλην των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο, αλλά ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σε μια άλλη παράγραφο λέει σε καμία περίπτωση να μην γίνει δεκτός κανένας τύπος χρηματοδότησης καμία απολύτως από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτό το τομέα. Κανένα είδος χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρωτοφανές. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα ε, μας ε, δυσαρεστήσει πια και τόσο πολύ αν μας λένε μη χρηματοδοτήσετε κάτι, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι ο μελλοντικό κοινοβουλευτικός έλεγχος, όπως λένε, για την πολιτική ασφάλειας, εξωτερική πολιτική, πολιτική άμυνας. η συμπεριφορά, η αντιμετώπιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι ότι είναι κακή ακριβώ η συμπεριφορά, αλλά λέει εντάξει, ποτέ όμως η καταστάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην γίνεται μια συνάντηση, να είναι πιο κατάλληλε οι εγκαταστάσει του Συμβουλίου που το ίδιο πολλές φορές μα ζητάει να χρησιμοποιεί τι δικές μας εγκαταστάσεις για συνεδριάσεις του Συμβουλίου, το ίδιο το Συμβούλιο. Λοιπόν, εδώ διαγράφονται δύο εναλλακτικές δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο ή μήπως να πούμε μία εναλλακτική. Τέλος πάντων, δύο λύσεις, μία πρόταση και μία εναλλακτική, αυτό θέλω να πω. Μια από τις δύο επιλογές είναι αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να δούμε πώς θα διαρθρώσουμε εν γέννη τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Τώρα να συνεχίσει η Κόζακ όπως ε, είναι σήμερα τα πράγματα, εντάξει, αλλά το να έχουμε εκπροσώπους 40 βουλών ουσιαστικά και εκπροσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα αντιμετωπίζονται έτσι με ποταπό τρόπο θα έλεγα και όταν έρχεται ο Μπαρόσο ή ο Φόνο Ρομπάι ε, απευθύνονται αποκλειστικά στους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί εμάς μας βλέπουν ε, συνέχεια. Ε, δηλαδή μας έχουν υποτιμήσει σαν να είμαστε ένα ξένο σώμα απέναντι στους ε, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σε ό,τι αφορά το τι γίνεται στην Κόζα και στι αρμοδιότητε, α μείνουν τα πράγματα ω έχουν. Αλλά σε ό,τι αφορά τι ευρύτερε, γενικές και πιο μόνιμες σχέσει μας, εγώ νομίζω ότι ή μπορούμε να πάμε σε ένα μηχανισμό ολοκλήρωσης ένταξης που από αριθμητικής και ποιοτικής πλευράς θα πρέπει να είναι διαφορετικό σε ό,τι αφορά το ένα εκπρόσωπος από τη μία πλευρά, 40 από την άλλη ή άλλη εναλλακτική που δεν με βρίσκει καθόλου να διαφωνώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα μου πείτε εσείς βέβαια. Δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια να συντονίζουν μεταξύ τους όπως θέλουν, να λένε ο ένας στο άλλο, το ένα στο άλλο ό,τι θέλουν, να έχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα διάφορα θεσμικά της όργανα μεταξύ αυτών και το Κοινοβούλιο όποια γνώμη και άποψη θέλουν και κάποια στιγμή, σε κάποια φάση της διαδικασίας, οι συντονίστρια αυτών των Εθνικών Κοινοβουλίων η αυτόνομη αυτή ε, αρχή, υπεύθυνη για τις πράξεις της, να συναντάται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επίσης για να συζητήσει, να καταλήξει συνενέσεις, και να συζητήσει παραλαμβάνω τα θέματα ε, για τα οποία έχουμε δεσμευθεί όπω προβλέπει η ίδια συνθήκη. Και εγώ νομίζω ότι αυτέ είναι οι δύο επιλογέ που έχουμε μπροστά μα. Και πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς δογματισμούς, χωρίς προκαταλήψεις. Όπως είπα, ένας μηχανισμός είναι να προχωρήσουμε σε μια ολοκλήρωση και δεύτερος δρόμος, πιο εύκολο για μας μονοπάτι αν θέλετε, εμείς φυσικά να συζητάμε, όπως είναι λογικό, για όλα τα θέματα, για οποιαδήποτε θέμα, με την αυτονομία και την υπευθυνότητα που έχουμε και τα Εθνικά Κοινοβούλια για λογαριασμό τους να συζητούν είτε σε μία γλώσσα, είτε σε δύο, είτε σε 21, να συνεδριάζουν, να εργάζονται, να συναντώνται όπου θέλουν, στην έδρα του, κοινοβουλίου, του Συμβουλίου συγγνώμη, ή σε κάποιο εθνικό κοινοβούλιο και όταν έρθει η στιγμή, μία φορά το χρόνο, δύο φορε το χρόνο, οπω συμφωνήσουμε τέλο πάντων, να συναντώνται μαζί μα για να συζητήσουμε για άλλα θέματα και πολιτική ασφάλεια, πολιτική άμυνα, εξωτερική πολιτική, να λέω ένα στιγμό, να λέω στη γνώμη του και τελικά να γίνει, να μην γίνει μια σύνθεση, αλλά όταν υπάρχει μια κριτική του ενός προς τον δεύτερο ή του δεύτερου προς τον ένα, να είναι μια λογική κριτική που να είναι κατανοητή. Δηλαδή να λέει κάποιο ότι δεν συμφωνώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να το εκφράζει. Και να λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν συμφωνώ με αυτό που λένε τα Εθνικά Κοινοβούλια και να το εκφράζει. Και να το αιτιολογεί. Αλλά όχι η σημερινή στάση τη ΚΟΖΑΚ που ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλου τομεί όπου συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά όπου μεγάλο μέρος του χρόνου του ουσιαστικά το, το καταναλώνει στο να ασκεί κριτική και να τιμωρεί κάποιες φορές αυτό το, το τμήμα της δικής του οντότητας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων που εκπροσωπείται επαξιότατα από τον πρόεδρο Καζίνη. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα ίσως είναι κάποιο είδους άσκηση πίεσης, ένα είδους lobbying προς τους ομολόγους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Για αυτούς που σιωπούν, αλλά έρχονται μετά να μας βρουν στο διάδρομο και να μας πούν ότι είναι αντίθετοι. Μα από τις ε, συνεδριάσεις δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή μόνο η ε, εχθρικότητα ε, τεσσάρων αλλά να φαίνεται και η στήριξη των 32. Αν έχουμε να αντιπαρατάξουμε όμως την εχθρική συμπεριφορά τεσσάρων και τη σιωπή, τη σιγή των υπολείπων, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και για την υπομονή που δείξατε ακούγοντάς με όλο αυτό το διάστημα και ελπίζω να, να καταλαβαίνετε την ειλικρίνεια με την οποία απευθύνομαι σε εσά. Γιατί δεν νομίζω ότι θα είχε καμία λογική ως συνάδελφοι να μην ε, μιλάμε με ειλικρίνεια, να μιλάμε τη σκέψη όπως μας έρχονται. Είμαι 12 χρόνια στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό και ήμουν 22 χρόνια στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχω καμία εχθρική στάση απέναντι στα Εθνικά Κοινοβούλια. Το αντίθετο. Δεν είμαι ένα ταλιμπάν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ένα εργαλείο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλο εργαλείο είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια και μπορούμε μαζί να συνεργαστούμε για να προοδεύσει η διαδικασία αυτή που είμαστε πολλοί από εμά αφιερωμένοι. Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μαρτίνες. Αυτά που μας είπες ε, δεν ε, ε, δεν σταμάτησαν στη μορφή. Μπήκαν στην ουσία και στο σχήμα, μπήκαν στην ουσία και όσον αφορά τι σχέσει ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις Εθνικές και τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, και κατ' επέκταση με την Επιτροπή και με τις αντίστοιχε κυβερνήσεις ε, εγώ έχω ακόμα την ε, αίσθηση που είχε η Επιτροπή μας στο Λονδίνο. Είχα σκοπό να σας μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Είχαμε λοιπόν μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας εδώ στην, ε, στο Λονδίνο. Ήρθαμε σε επαφή με τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου καθώς επίσης και τον υπεύθυνο, τον επικεφαλής μάλλον της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των, της Βουλής των Λόρδων και πρέπει να σας πω ότι ειδικά στην πρωινή συνεδρίαση η αντιπαράθεση ήταν σημαντική διότι κατέστη σαφέστατη η εχθρικότητα ε, της, ε, των οργάνων αυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέρα από την συνάντηση που είχαμε ε, με την Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων της Βουλής των Λόρδων ε, που τα πράγματα ήταν λίγο πιο καλά ε, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις είχαμε πολύ αρνητική στάση. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της συνθήκης της Λισαβόνας, οποιαδήποτε περαιτέρω αρμοδιότητα θα μπορούσε να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έπρεπε να γίνει μέσα από συνεμαντική νομοθετική διαδικασία το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, επομένως καταλαβαίνουμε ότι εμείς δεχτήκαμε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν είναι ένα πέρασμα προς κάτι ακόμα πιο πέρα. Είναι το μεγαλύτερο, το μέγιστο που θα μπορούσαμε να δεχτούμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ε, το κοινοβούλιο του Πρωθυπουργού Κάμερον θα δέχεται εντολές κατά κάποιο τρόπο από άλλα κοινοβούλια. Με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την πραγματικότητα λοιπόν θα πρέπει να λογαριαστούμε. Νομίζω λοιπόν και είναι η προσωπική μου εντύπωση η οποία σχηματίζεται σιγά σιγά είναι λοιπόν η προσωπική μου εντύπωση ότι ο χώρος τον οποίον ε, δημιουργείται η καλύτερη ολοκλήρωση της Ευρώπης, αυτό το φόρουμ είναι η ΚΟΖΑΚ. Και επομένως βεβαίως δεν υπάρχει λόγος να συνεδριάζουμε μια φορά στα τόσα ε, θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης, State of the Union. Και Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που οι ύπατοι αξιωματούχοι, Μπαρόζο και Βαν Ρόμπε, ήταν παρόντες γιατί νομίζω ότι παλιότερα δεν ε, ε, είχαμε τόσο σημαντικούς συμμετέχοντες. Ε, και σίγουρα θα έχουμε και στην επόμενη συνεδρίαση είτε τον ίδιο τον Μπαρόζο είτε τον Σεύκοβιτς και σίγουρα θα υπάρχει και ο Ούγγρος Υπουργός. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό το μήνυμα που στέλνουμε ε, και προς, προς τους πολίτες της Ευρώπης γιατί καλό είναι που τους λέμε θα πρέπει να γίνουν ζυμώσεις, θα πρέπει να συμμετάσχετε και εσείς στις ζυμώσεις αυτές αλλά εάν ε, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι μας δεν συμμετέχουν τότε πώς θα πείσουμε Ε, και ξέρετε εγώ βλέπω το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όπως είναι τα δύο κοινοβουλευτικά όργανα κάποιων χωρών. Όπως υπάρχει άνω κάτω Βουλή, υπάρχει ε, το Κοινοβούλιο των Κρατών που είναι το Συμβούλιο και υπάρχει ε, και το Κοινοβούλιο των Λαών που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε τις εργασίες μας στην Επιτροπή μας σκεπτόμενοι την απόφαση της 30ης Ιουνίου 2008 ε, που, ήταν, που έθετε και κάποιους όρους κατά κάποιο τρόπο στο οικοδόμημα της ε, Ευρώπης αλλά ε, πιστεύω ότι σε αυτήν την διάσταση της επικοινωνίας της Ευρώπης θα πρέπει να συμμετάσχει κατά κάποιο τρόπο και η ΚΟΖΑΚ Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, διάφορα σημεία στα οποία ενδεχομένως έχουμε υπερβάλλει. Έχουμε εδώ και τον συνάδελφο Άντζελ. Ε, ενδεχομένως ε, επιμείναμε πολύ έτσι ώστε να υπάρχει παρουσία του Κοινοβουλίου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος των λαών και δεν είναι δυνατόν να έχουμε εκπροσώπους 40 κοινοβουλίων ε, Γκουερέρο έχει ζητήσει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνεφ για τις πληροφορίες και για την ανάλυση κυρίως που μας ε, έκανε. Είναι γεγονός ότι ε, εντάξει χρόνια πολλά μεν για τα γενεθλιά σας αλλά αν λάβω υπόψη όλες τις αρμοδιότητες που έχετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, φαντάζομαι ότι πρέπει να είστε σε τέλεια φόρμα και φυσική κατάσταση. Αυτό πρέπει να σας ευχηθούμε για να συνεχίσετε να φέρετε σε πέρα στα καθήκοντά σας. Σε ό,τι αφορά τώρα μια συγκεκριμένη συνεδρίαση των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, η περιγραφή που μας έκανε αυτή τη συνάντηση ο κύριος θα νομίζω αποτελεί διάγνωση των, ε, της κατάστασης και των σχέσεων. Δεν είναι η αφήγηση κατά η περιγραφή των σχέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά είναι περιγραφή των αδρών γραμμών, των σχέσεων μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, που μας ανησυχούν και για το μέλλον ε, του Ευρωπαϊκού Οικοδόμητος και για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας είπε ο πρόεδρος Κασίνη ότι στην επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο εκεί είδε σε ποιο, ως ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η ιδέα ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι ένα βήμα παραπέρα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, αλλά είναι το τελευταίο σημείο, είναι ο τερματισμός. Το σημείο του τερματισμού. Δηλαδή ε, ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη δυναμική υπαναχώρησης. Δηλαδή δεν θεωρείται ε, ένα σημείο στο οποίο φτάσαμε ένα σημείο τερματισμού η συνθήκε της Λισαβόνας αλλά ένα σημείο στο οποίο δεν έπρεπε να είχαμε φτάσει. Δηλαδή, ε, μιλάμε για κάτι χειρότερο από απλή παράλυση της κατάστασης στην οποία είχαμε φτάσει με τη συνδέκη της Λισαβόνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, εγώ, ε, σε αντίθεση με τον κύριο Μαρτίνο που είναι 12 ε, χρόνια ευρωβουλευτής και 22 βουλευτής ε, στο Εθνικό, Κοινοβούλιο, εγώ για πρώτη φορά είμαι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και ποτέ δεν υπήρξα εθνικός βουλευτής. Νομίζω ότι η προηγούμενη φάση όπου ο ευρωβουλευτή ήταν και εθνικό βουλευτής, δημιουργούσε, ε, μάλλον προκαλούσε λιγότερες αντιστάσεις από πλευρά εθνικών βουλευτών απέναντι στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σίγουρα αυτό είναι μεγάλη πρόοδος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να είναι κάποιος ευρωβουλευτής Ω κάτι ξεχωριστό. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό δημιούργησε αντιδράσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια και δημιούργησε αντιστάσεις, το είπε και ο κύριο Μαρτίνεθ, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου. Για πολύ καιρό, πολλοί εθνικοί βουλευτέ έβλεπαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μια βουλή αποκλειστικά για συζήτηση, για μελέτες, για προβληματισμό, για παρουσίαση και υποβολή προτάσεων δεν καταλάβαιναν ότι επηρέαζε τον ρόλο ε, ε, των, αρμοδιοτήτων της εξουσίας που είχαν στα εθνικά κοινοβούλια. Και τώρα που αυξάνονται οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυστυχώς αρχίζουν οι εθνικοί βουλευτές να το βλέπουν ως ανταγωνιστή και όχι ως ένα σώμα, ένα φόρα με τον οποίο πρέπει να συντονιστούν. Επίσης, σε ό,τι αφορά την, κρά, την επανεθνικοποίηση κάποιων πολιτικών ή τάση μάλλον, αν ε, προτιμάτε τον όρο, τάση επανακρατικοποίησης κάποιων πολιτικών. Αν δηλαδή κάποιες πολιτικές ευρωπαϊκές διάστασεις θα έπρεπε να γυρίσουν πίσω και να γίνουν εθνική αρμοδιότητα. Παραδείγματο χάρη, συζητήσει για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση είδαμε πόσο πολύ ε, αντιστάθηκαν πολλές χώρες και πολλά, πολλές εθνικές οργανώσεις σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς χρηματοοικονομικής εποπτείας, οικονομικής διακυβέρνησης, πόσο αντιστάθηκαν στο να έχουν αυτοί οι οργανισμοί, επαναλαμβάνω, μια ευρωπαϊκή ε, ταυτότητα, ένα ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Επίσης, ε, Αντίθετα λειτουργεί και μία τάση που βλέπουμε λιγότερο σε κάποιες άλλες χώρες και περισσότερο σε κάποιες άλλες, ότι δηλαδή σε περίοδο κρίσης βλέπουμε ένα είδος ε, δαιμονοποίησης των ε, Βρυξελών για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Σε αυτή την ιστορική περίοδο είναι αποφάσεις ε, που έχουν να κάνουν με περιορισμούς, με περικοπές του προπολογισμού, με μείωση των κοινωνικών πολιτικών. Ε, πολλές φορές σχετίζονται με το πρόβλημα της ανεργίας και σε πολλές χώρες ε, οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις για να προστατευθούν εξηγούν ότι ίσως οι ίδιες δεν θα υποστήριζαν αυτά τα μέτρα αλλά τους τα επιβάλλουν οι Βρυξέλλες, αυτή η υπερδομή που κανείς ε, δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι ή που είναι, αλλά την ταυτοποιούν με τις Βρυξέλλες, την ταυτίζουν με τις Βρυξέλλες. Κατηγορούνται οι Βρυξέλλες λοιπόν. Δεν ξέρω αν ξέρετε και την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστήριου που πέραν των ερμηνειών επί της ουσίας ε, είναι συμπαθής και αρεστή σε πολλούς πολίτες, κυβερνήσεις, φορείς, ε, κοινοβούλια. Μπορούν να σκεφτούν δηλαδή ότι τελικά πήγε υπερβολικά μακριά η ευρωπαϊκή οικοδόμηση και αρνούνται, όπως και η απόφαση αυτή, τουλάχιστον ε, αν όχι ε, αρνείται, ξεχάστε τη λέξη αρνείται, θέτει υποαφισβήτηση αμφιβάλλει για την πλήρη δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε λοιπόν σε μια ιστορική χρονική στιγμή όπου ξανά μιλάμε για έθνη κράτη, για τους φορείς και τους οργανισμούς των εθνικών κρατών που είναι η βάση οικοδόμησης του ευρωπαϊκού σχεδίου και ό,τι έχει προσθεθεί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, κοινοτικοποίηση πολιτικών κτλ. κτλ αυτά όλα ε, τα αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Υπό την έννοια αυτή, οι προτάσεις του κ. Μαρτίνεθ και πλησιάζω στην ολοκλήρωση της παρέμβασής μου, νομίζω ότι μας ε, δημιουργούν την πρόκληση στην Επιτροπή μας, συγκεκριμένα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά, την πρόκληση να ξαναχτίσουμε την ευρωπαϊκή αυτή ορμή, εξηγώντας ότι είναι ένα σχέδιο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα έλεγα. Έχουμε το ευρωπαϊκό, έχουμε το εθνικό, έχουμε το περιφερειακό επίπεδο. Και υπάρχουν και χώρες που έχουν έτσι αναπτυγμένο αυτό το περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μπορούμε να έχουμε λοιπόν και μία φάση συνεργασίας ή μία φάση αντιπαράθεση. Η φάση αντιπαραθεση αποδυναμώνει όλα τα επίπεδα. Αποδυναμώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποδυναμώνει τα εθνικά κοινοβούλια και βέβαια αποδυναμώνει και τα περιφερειακού τύπου κοινοβούλια. Όταν το καθένα αγωνίζεται να κρατήσει ή να έχει αρμοδιότητες που ασκούνται από κοινού κανονικά, ποιο είναι το συμπέρασμα που μπορούμε να συναγάγουμε από αυτό, είναι ότι η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση είναι αυτή οι οποία Και τα εθνικά κοινοβούλια πλήττονται. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια όμως πρέπει να ασκούν τις νομοθετικές του αρμοδιότητες και τον έλεγχο που τους ε, αναγνωρίζουν οι διατάξεις και οι συνθήκες. Τώρα, Έχουμε κάποια πολιτικά κόμματα της ίδιας ιδεολογικής οικογένειας σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχει ένα κοινό σχέδιο. Υπάρχει το πολιτικό, το θεσμικό επίπεδο σε αυτό το σχέδιο και υπάρχει και το επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Όλοι μαζί πρέπει να εργαστούμε γιατί αλλιώς το αποδυναμώνουμε όλο αυτό το οικοδόμημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μέσερ Σμιτ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον, τον συνάδελφο για την ε, εισήγησή του. Συμφωνώ για πολλές, σε πολλές από τις ε, περιγραφές της κατάστασης. Να πω ωστόσο ότι θεωρώ ότι όλοι όσοι έχουν δημόσια θέση και ασκούν δημόσιο λειτουργίαμα το κάνουν αυτό με τις καλύτερες των προθέσεων. Και όταν ξεκινάμε διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Άρα, μας υποχρεώνει η συνθήκη της Λισαβόνας να κάνουμε το έργο αυτό. Άρα, θεωρώ ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μπούμε και να δούμε ε, πώς θεωρούν την κατάσταση όσοι είναι εχθρικοί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν περιορίζεται στους Φιλανδούς, στους Βρετανούς και στα σχετικά κοινοβούλια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ίσως να μην υπάρχει εχθρότητα, αλλά υπάρχει, ξέρετε, μια επιφυλακτική στάση, ένας σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Κοιτώντας λοιπόν τις εξελίξεις του τελευταίου χρόνου, του τελευταίου 1,5 χρόνου από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν είναι δύσκολο να βρούμε τα όπλα μας. Για παράδειγμα το EAS. Πού ήταν πριν από 1,5 χρόνο και πού είναι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαπραγματεύτηκε τον ε, προϋπολογισμό και κάποια από τα θέματα αυτά, κάποιε από τι αρμοδιότητε, εγχωρήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Επιτροπή. Κάποιε από τι αρμοδιότητε που ήταν στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ευρωπαϊκής ε, πλευράς, από πλευράς Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Φυσικά αυτό είναι εύλογο γιατί ε, διαπραγματευόμαστε, συζητούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ούτω καθεξής. Από εθνική όμως προοπτική μπορεί να θεωρηθεί ως ε, μία υπόσχεση που αθλήθηκε. Και πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, να αντιληφθούμε την πραγματικότητα αυτή καθώς συμμετέχουμε στην απόφαση αυτή και όταν μιλάμε για υποχρέωση εκπλήρωση των καθηκόντων μας θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί κάποια εθνικά κοινοβούλια βρίσκονται αυτόματα σε μια θέση πιο εχθρική ένατη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν κάποια πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι κοιτάξτε δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ αυτό γιατί δεν καταλαβαίνετε τίποτα και θα σας εξηγήσουμε εμείς πώς έχουν τα πράγματα. Αυτό το μόνο που θα καταφέρει είναι να δημιουργήσει πιο πολύ εχθρική στάση. Ή μπορούμε να πούμε, ωραία, ας κάνουμε τη συζήτηση αυτή, ας ανοίξουμε τα έγγραφα αυτά και αυτό κάνουμε στο Κόζακ. Με μεγάλο δισταγμό παρευρέθηκα στην τελευταία συνάντηση, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια συζήτηση. Γιατί ξέρετε κάποιοι, χάρη στη σωστή επιχειρηματολογία, άλλαξαν ακόμα και τη θέση τους, άλλαξαν ακόμα και την ψήφο τους. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την ανοιχτή συζήτηση. Αντί να προσπαθούμε να αποδείξουμε στους ε, αντιπάλους μας ότι έχουν λάθος και κάνουν λάθος, ας τους το τεκμηριώσουμε, ας τους το αποδείξουμε. Να τους το καταδείξουμε, να επιμείνουμε στον πρόεδρο της ΚΟΖΑΚ ότι μέχρι ότου πετύχουμε συμφωνία για τον έλεγχο στα πλαίσια του ΕΕΣ σε ό,τι αφορά την αρχή της επικουρικότητας, δεν θα μπορέσει να υπάρξει συνάντηση ΚΟΖΑΚ χωρίς τέτοια ατζέντα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαθεσμική συμφωνία που θα τα ρυθμίζει αυτά. Και δεν βλέπω να υπάρχει άλλη εναλλακτική πέρα από το να επιμείνουμε και τελικά να πετύχουμε να επιληθούν οι παρανοήσεις οι οποίες προφανώς υφίστανται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Σόνεγκαρντ. Øh, øh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την, ε, αν μη τι άλλο, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αναφερθήκαμε εντελεχώς λοιπόν στην κατάσταση έτσι όπως αυτή έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Νομίζω πως η ανάλυση είναι ορθή. Και είναι γεγονός ότι σε μερικά κοινοβούλια βλέπουμε πολύ επιθετική στάση απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ερώτημα ε, που πρέπει να θέσουμε σε αυτούς είναι το εξής. Γιατί συμβαίνει αυτό. Τι εκφράζεται μέσω αυτής της στάσης. Και μπορούμε να το δούμε σαν ένα κύκλο στο εσωτερικό του οποίου βλέπουμε το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια με τις αντιθέσεις τους και με τις διαφορές τους. Νομίζω ότι άλλωστε αυτό καταδεικνύει μια ε, ε, ευρία τάση και κατά αυτή την έννοια αποτελεί και ένα ευρύ πρόβλημα. Και στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει την αντίδραση των λαών απέναντι στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι απαραίτητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει για υπερβολικά πολλά πράγματα. Μεγάλος αριθμός των ψηφοφόρων μας δεν πιστεύει πλέον σε αυτά που λέμε και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε το ένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε το άλλο και δεν κάνει διαφοροποίηση μεταξύ του Συμβουλίου, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η, η γενική αίσθηση λοιπόν του κόσμου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει υπερβολικά πολλές αποφάσεις για υπερβολικά πολλά θέματα και ακριβώς με τον τρόπο αυτό οδηγούνται κάποια κοινοβούλια, εθνικά κοινοβούλια, σε αυτή την εθνική στάση απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε λοιπόν να τους πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κατά κάποιο τρόπο το θύμα αυτής της έλλειψης ικανοποίησης του κόσμου, των πολιτών της Ευρώπης. Και στο ερώτημα πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει για υπερβολικά πολλά πράγματα. Ισχύει αυτό. Πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν ε, μήπως πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα την κατάσταση στους πολίτες έτσι ώστε να μην έχουν πλέον αυτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει για υπερβολικά πολλά πράγματα. Ο κύριος Μαρτίνες αναφέρθηκε σε διάφορα σκανδιναβικά κοινοβούλια και καταλαβαίνω γιατί. Γιατί στη Σκανδιναβία είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το βάζουν εντό εισαγωγικών γιατί έτσι το λένε κιόλα, έτσι το βλέπουν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ε, πήρε αποφάσεις ε, ε, Ε, είχαμε και μία σειρά αποφάσεις όπως η Viking Line, η Vaxol, ε, αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αποφάσεις οι οποίες είχαν μεγάλη επίπτωση και στη Σουηδία και στη Δανία και στη Φιλανδία. Οδήγησε σε μείωση των δικαιωμάτων τους και επομένως δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες των χωρών αυτών γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχωσε τη μύτη της και ε, άλλαξε κάποια πράγματα. Στη Δανία άλλαξε το σύστημα των συλλογικών συμβάσεων μετά από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου που αποφάσισε ότι δεν είχαμε δικαίωμα να απαιτούμε ε, ότι οι Πολωνοί εργάτες ή οι Πολωνοί εργαζόμενοι ε, που έρχονται στη Δανία δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Δανέζους εργαζόμενους. Και όμως αυτή είναι η απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Βεβαίως το Κοινοβούλιο έπαιξε θετικό ρόλο όταν η Κομισιόν αποφάσισε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να δεχτούν ε, κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε για το κρέας. Δεν ξέρω τι έγινε στην ε, Ισπανία, αλλά καμία χώρα από τις σκανδιναβικές χώρες δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι θα πρότεινε κάποια στιγμή να γίνεται αποδεκτή μια τέτοια ουσία στο κρέας. Ε, και όμως κάποια στιγμή το, το, η Κομισιόν είπε ορίστε δεχόμαστε πλέον αυτή την ουσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως υπάρχει λόγος που οι πολίτες εκφράζουν αυτή την επιθετικότητα. Υπάρχει λόγος που τα κοινοβούλια εκφράζοντας αυτήν την απέχθεια ας πούμε ε, ε λειτουργούν με αυτόν τον ενετικό τρόπο. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά βεβαίως δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται μονάχα στις συνεδριάσεις της ΚΟΖΑΚ. Για να, αντικρούσουμε όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει οπωσδήποτε να τα συζητήσουμε πρώτα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ραντζέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να πω. Με μεγάλη προσοχή την ε, παρουσίαση του φίλου μας, του συναδέλφου Μαρτίνες, αλλά θα πρέπει να πω, μάλλον να παραθέσω μία πρόταση από τη βίβλο «Ουδέ νεότερον υπό τον ήλιο». Γιατί μετά την επικύρωση της της Λισαβόνας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, βλέπουμε την πολιτική σχέση μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χαρακτηρίζεται από μια θεσμική, θα έλεγα, ζήλια. Και θα πρέπει να πω ότι είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι στο σημείο αυτό από πλευράς εθνικών κοινοβουλίων υπάρχει μια στάση εσφαλμένης προπτικής. Και αυτό το λέω χωρίς να φοβάμαι τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Είναι σφάλμα. Επειδή πιστεύω και είμαι πεπισμένος, επίσης, ότι το Συμβούλιο μέσω της διακυβέρνησης τους που συνήθως υποστηρίζει το Κοινοβούλιο, προσπαθεί να κάνει μια εκστρατεία να πείσει τα εθνικά κοινοβούλια ότι μετά τη θέση σε εφαρμογή της Λισαβόνας θα χάσουν κάποιες αρμοδιότητες, κάποιες εξουσίες τις οποίες θα εκορυθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε το επιχείρημα αυτό το οποίο άκουσα και να το δούμε, να δούμε πόσο ευθύνεται για τη σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί ακούγεται συχνά, χιλιάδε φορέ το έχω ακούσει, ότι ελέγχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όχι μόνο υποστηρίζω την άποψη του συναδέλφου Μαρτίνε, αλλά και ω μέλο Εθνικού Κοινοβουλίου και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας έχω δει ότι δεν είναι πολύ απλό να ελέγχει το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο την κυβέρνησή του. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι το Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί να ελέγξει, δεν μπορεί να ελέγξει, δεν μπορεί να ελέγξει τις άλλες 26 κυβερνήσεις που είναι στο Συμβούλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούν να ελέγξουν την θέση του Κοινοβουλίου εκτός και αν υπάρχει ρήτρα ομοφωνίας. Τότε μόνο υπάρχει μια δυνατότητα ελέγχου της θέση του Συμβουλίου. Ιδάλω δεν υπάρχει δυνατότητα γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τον Συμβούλιο. Όχι, ελέγχουν μία κυβέρνηση. Ένα μόνο κυβερνητικό σχήμα μεταξύ των 27. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έλεγχος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με διαφορετικό τρόπο και του Συμβουλίου mm. και τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουν. Mm. Φυσικά, εγώ πιστεύω και συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο με αυτά που μας ανέφερε ο συνάδελφος Σμιτ ο οποίος ανέφερε ότι ιδιαίτερα στην ΚΟΖΑΚ, δηλαδή όταν έχουμε και τις 27, και τους 27 εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί αυτή η θέση. Ανεκτά, θα έλεγα, χωρίς ε, φόβο. Χωρίς φόβο παρανοήσεων. Ειλικρινά όμως πιστεύω και αυτό μου το υπαγορεύει η εμπειρία μου, ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε και τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάθε Εθνικής Βουλής ή όπως είπε ο συνάδελφος Μαρτίνης Μαρτίνες με καινοτομικό τρόπο το παρουσίασε τι σχέσει με τα εθνικά κοινοβούλια που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο γιατί ακόμα και σε χώρε χωρίς ομοσπονδιακό καθεστώς υπάρχουν περιφερειακά κοινοβούλια με τις ε, δικές τους αρμοδιότητες. Άρα με το συνοφίλευμα εθνικών κοινοβουλίων θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση σχέση και πρόσφατη ήταν η εμπειρία που είχα με την αντιπροσωπεία την, της οποίας προέδρευσε ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, ο κάλο Καζίνη, στο Λονδίνο όπου πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι συζητούσαμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το νομοσχέδιο για τις ευρωπαϊκούς προθεσμούς, είδα και αντιαισθάνθηκα μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, δεκτική προς την άποψή μας. Όχι ότι τη δέχτηκαν την άποψή μας, αλλά τη συζήτησαν. Έδειξαν ανοιχτό πνεύμα και δεκτικότητα. Και θεωρώ ότι τέτοιε διμερεί σχέσει πρέπει να αναπτύξουμε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Εθνικού, των Εθνικών Κοινοβουλίων, μεμονωμένων. Όχι μόνο σε τέτοια μορφή και με τα 27 κοινοβούλια μαζί να υπάρχει και διμερής επαφή, γιατί πολύ απλά είναι πιο απλό να εξηγήσουμε, να συζητήσουμε με ειλικρίνεια και ανοιχτό πνεύμα έχουμε αρκετό χρόνο να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας και δεν υπάρχει αυτή η εκστρατεία, ξέρετε, δεν υπάρχουν ε, αυτή η τάση να διακρίνεται ένα εθνικό κοινοβούλιο όπως το Φιλανδικό Κοινοβούλιο και μετά να θέλουν όλοι να δεχθούν σε πρωταθλητές για να αποδείξουν ότι είναι οι πιο καλοί ε, βουλευτές, ότι είναι πιο καλή από τους άλλους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ήταν στη Βουλή των Λόρδων, μας ρώτησαν για παράδειγμα για κάποια θέματα, ιδιαίτερα ένα θέμα το οποίο έθεσε και το Φιλανδικό Κοινοβούλιο, το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι μετά από κάποια συζήτηση και ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι είδαμε ότι οι βουλευτές ήταν σαφώς ενημερωμένοι για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, κάτι το οποίο δεν ε, ε, συμβαίνει πάντα, εξαρτάται από το Κοινοβούλιο. Όχι, στην Βουλή των Λόρδων είναι πάρα πολύ ακριβείς και γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει μετά τις εξηγήσει που δόθησαν λοιπόν, που τους δώσαμε. Είδα μια ατμόσφαιρα και ένα πνεύμα δεκτικό. Μας κατάλαβαν. Φυσικά, θα πρέπει να βρεθεί μια θεσμική λύση. Για την Κόζακ, και τα σχετικά ζητήματα θα πρέπει να βρεθεί μια θεσμική λύση και συμφωνώ με τις λύσεις που μας παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος Μαρτίνες Μαρτίνες και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση δημοσίων σχέσεων σε ό,τι αφορά το διμερές επίπεδο. Είναι εντελώς διαφορετικό είναι εντελώς διαφορετικό πώς αντιμετωπίζονται οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μία διμερή, επαφή σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται σε μία κοινοβουλευτική συνάντηση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε θεωρώ και θα πρέπει να το κάνουμε μάλιστα ως προληπτική στρατηγική γιατί πολλά κοινοβούλια και πολλοί βουλευτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά ζητήματα θεωρώ ότι αν διαθέτουν όσες πληροφορίες χρειάζονται ασφαλώς και θα σχηματίζουν πάντα τη δική τους άποψη και αυτό είναι εύλογο και θεμητό αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα ξεκινούν το διάλογο χωρίς προκαταλήψεις εναντίον μας. Και για να κλείσω θα ήθελα να τονίσω ότι είμαι πεπισμένος ότι εδώ ε, υπάρχει έντονη επιλογή από πλευρά του Συμβουλίου. Πέρα από την υποστήριξη κομμάτων, σε κάποιες περιπτώσεις υποστηρίζονται και ομάδες του Κοινοβουλίου, αλλά μέσω εθνικού επίπεδου και αυτό το είδα και μετά τις διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας Πλαισίου, γιατί ήταν σαφές πλέον ότι υπήρξε παρανόηση, παραπληροφόρηση. Στοχευμένη παραπληροφόρηση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αυτό το είδαμε και στη Βουλή των Λόρδων. Γιατί όταν ξεκινήσαμε και αρχίσαμε να εξηγούμε, όπως είπε ο κ. Καζίνη, ότι στη διεθνή διάσταση μπορούμε να πούμε ότι το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό έχασε σε όλα τα μέτωπα, ότι τα πράγματα έμειναν λίγο πολύ όπως είχαν πριν από τη Συμφωνία Πλαίσιο και ότι δεν ε, πέρασαν ουσιαστικά ε, ιδιαίτερε αλλαγέ και ότι σε άλλα ζητήματα υπήρξε ουσιαστική πρόοδο, μα είπαν ότι εντάξει. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δεν έγινε τίποτε, δεν άλλαξε τίποτε ουσιώδες, τίποτε νευραλγικό στα θέματα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η διμερής στρατηγική όπου έκανε πολύ σημαντική δουλειά και η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σε ό,τι αφορά και τις ε, επισκέψεις μας στις διάφορες πρωτεύουσες. Θεωρώ ότι μπορεί να έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Συναντηθήκαμε λοιπόν και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο, τουλάχιστον εγώ σε αυτές τις αντιπροσωπείες ε, συμμετείχα, συναντήσαμε λοιπόν τα μέλη τα οποία ε, κανονικά συμμετέχουν στην ΚΟΖΑΚ. Και αυτό φυσικά ήταν πάρα πολύ καλό γιατί είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Θα έλεγα σχεδόν να πείσουμε, θα αποφύγω όμως τον όρο, να συζητήσουμε τα θέματά μας και να εξηγήσουμε τις δικές μας θέσεις. Ευχαριστώ πολύ και για την αισιοδοξία που εκφράσατε. Ήπιος όμως, μετριοπαθής ε, η αισιοδοξία μου. Ναι, ναι, γιατί είστε και λογικός. Ναι, πρέπει να δούμε τα, ε, να βλέπουμε κατάματα και τις ε, δυσκολίες, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε σε αυτή την οδό. Και πιστεύω ότι σωστό είναι και καλά κάνατε και υπογραμμίσατε τη σημασία των διμερών σχέσεων γιατί καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα, γιατί λύνονται προβλήματα κτλ. Σέφλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μαρτίνες. Εξαιρετική συζήτηση. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα θέμα εξουσίας. οι εξουσίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέρχονται από άμεσες εκλογές, αλλά τα εθνικά κοινοβούλια και μέσω εγχωρίων πολιτικών διαδικασιών ε, επιβεβαιώνονται οι εξουσίες ε, των άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν έτσι μια, μια διάσταση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο, ολοένα και αυξανόμενος ε, ρόλος του Κοινοβουλίου, οι ολοένα και αυξανόμενες εξουσίες του και θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Έχουν αλλάξει λοιπόν κάποια πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν αυτές τις αλλαγές. Ε, ξαφνικά ε, τα εθνικά κοινοβούλια ξύπνησαν και είπαν «Α, για δες, τα πράγματα είναι έτσι». Λες και δεν το ήξεραν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Η Κόζακ και η στάση κάποιων στην Κόζακ είναι σύμπτωμα ε, μιας γενικότερης ασθένειας. Και δεν είναι ίσως πολύ κακό που το πρόβλημα αυτό αναδύθηκε στην Κόζακ, όπου που είναι ένα φόρουμ κατά την άποψή μου μπορούν να συζητηθούν ε, τα θέματα αυτά. Ένα από τα προβλήματα τα οποία θεωρώ εγώ σημαντικά ε, είναι ότι ε, σε πολλές περιπτώσεις είμαστε το μεγάλο ερωτηματικό ε, για τους πολίτες αλλά και για τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν ξέρουν τι κάνουμε ακριβώς. Επομένως, ε, ναι μεν προκαλούμε την ε, περιέργειά τους. Και ξέρετε, εγώ έχω έρθει σε επαφή κάποια φορά με εθνικούς βουλευτές και μου λένε «Μα τι ακριβώς κάνετε, τι μαγειρεύετε εκεί που είσαστε εσείς». Και σε πολλές περιπτώσεις ε, ε, με την ε, βοήθεια και των εθνικών κυβερνήσεων, τα εθνικά κοινοβούλια δημιουργούν την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει παραπάνω από αυτά που πρέπει και ότι ξεπερνάει τα εσκαμμένα όσον αφορά κάποιες αποφάσεις. Επομένως, χρειαζόμαστε καλύτερη επικοινωνία. Πιστεύω ότι πραγματικά ό,τι και αν πιστεύει κανείς και όποια και είναι η φιλοσοφική του προσέγγιση του θέματος της επικοινωνίας, πιστεύω ότι η πληροφόρηση, η επικοινωνία είναι αυτή που χρειάζεται. Καλύτερη, περισσότερη πληροφόρηση έτσι ώστε οι τοπικέ κυβερνήσει, οι περιφερειακέ κυβερνήσει, οι κεντρικέ κυβερνήσει, τα τοπικά κοινοβούλια, τα περιφερειακά, τα εθνικά να ε, κατανοούν ακριβώ περί τίνο πρόκειται, να μα ξέρουν, να ξέρουν τι κάνουμε. Και κατά αυτή την έννοια, οι διμερεί συναντήσει, πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσει, είναι καλέ. Βεβαίως λοιπόν μπορούμε να έχουμε όλο και περισσότερες ε, ε, διμερείς ε, συζητήσεις. Δεν ήμουν παρόν στη συναντήση στο Λονδίνο, αλλά ε, μπορώ να καταλάβω πολύ καλά το κλίμα που περιγράφεται. Επίσης, στο τρίο των Προεδριών υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν έτσι ώστε η αναγνωρισιμότητα του έργου του Κοινοβουλίου να γίνει πιο σαφής. Δεν έχουν γίνει αρκετά βήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω, μάλλον να συγχαρώ και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Αντιπρόεδρο. Εγώ στη Γερμανία συχνά βλέπω ότι μεταξύ των ομόσπονδών κρατηδίων και μεταξύ του Εθνικού Κοινοβουλίου υπάρχει η συζήτηση αυτή την οποία κάνουμε και εδώ ε, το ποιο είναι αρμόδιο γιατί και πράγματι το θέμα είναι παιχνίδι εξουσία Θεωρώ όμω ότι τα κοινοβούλια σε εθνικό επίπεδο αλλά και τα περιφερειακά κοινοβούλια είναι σύμμαχοί μας ουσιαστικοί και αυτό θα πρέπει να το, ε, να το αναγνωρίσουμε και να βρούμε μέσα για τη βελτίωση της συνεργασίας αυτής στο γερμανικό Bundestag μετά από δύο χρόνια νομίζω άνοιξε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες όπου, εκπρε, όπου εκπροσωπούνται όλες οι, όλα τα κόμματα και όλοι γνωρίζουν ότι έχουν ένα άτομο επαφής γιατί ε, εν μέρη δεν τους ε, ενημέρωνε επαρκώς η κυβέρνησή τους. Και αυτό ήταν ο λόγος ε, για τον οποίο οι εθνικοί βουλευτές της Γερμανίας αποτάνθηκαν στο συνταγματικό δικαστήριο και κατηγγείλαν την συνθήκη της Λισαβόνας και το συνταγματικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εφαρμογή δεν είπαν ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι σωστή, αλλά ότι η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο δεν ε, εγγυάται τη συμμετοχή του, του Γερμανικού Κοινοβουλίου που θα έπρεπε να υπάρχει. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα μέσα συνεργασίας και στις ε, πρωτεύουσε και αυτό το ζητώ από το Προεδρείο να δούμε τι μέσα μπορούμε να παρέχουμε αν ένας βουλευτής ε, Εθνικού Κοινοβουλίου επεξεργάζεται ένα θέμα το οποίο, στο οποίο μπορούμε να τον βοηθήσουμε και με το οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή με ένα γραφείο επαφή, γιατί το θέμα αυτό το πραγματεύεται και ένα ε, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Ζόντρ, κάτι και εσεί το είπατε αυτό. Είναι πάντα κακό να λαμβάνουν πολιτικέ αποφάσει στα δικαστήρια, ξέρετε. Και αυτό το ισχύει και για το εθνικό επίπεδο. Όχι. Όταν λαμβάνουν αποφάσεις ε, τα δικαστήρια, δημιουργείται ένα κενό αέρα και δεν υπάρχουν ε, νόμοι. Όχι, θα πρέπει λοιπόν ως συμμάχους να τους αντιμετωπίζουμε τους ε, βουλευτές και να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο. Γιατί στο Συμβούλιο, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι όλοι πολιτικοί εσωτερικών και ασκούν πολιτική εσωτερικών στο Συμβούλιο. Και ξέρετε τι γίνεται το συνεδριάσει το Συμβούλιο. Όλα γίνονται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική μας, υπόσχονται ότι οι συμβιβασμοί θα κρατήσουν και ο κάθε υπουργό φτάνει στην χώρα του και λέει καταφέραμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Είναι σαφές αυτό και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής μας για το πώς θα συνεργαστούμε καλύτερα με τους συμμάχους μας, τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και ο κύριος Καζίνη ήταν ε, πρόεδρος της Επιτροπής της ε, Αντιπροσωπείας στο Βερολίνο. Να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ καλές οι εντυπώσεις από το γεγονός ότι χρησιμοποίησατε και αφιερώσατε χρόνο στους εθνικούς βουλευτές και να δούμε και τι θα γίνει και σε πλευρά υπαλλήλων. Ίσως από τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να έρθουν βοηθοί και να τους υποδεχτούμε με ανοιχτή αγκαλιά για να μάθουν πώς λειτουργούμε, να καταλάβουν και ξέρετε είναι και το γλωσσικό εμπόδιο γιατί εμείς το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και το αμελούμε ίσως, αλλά υπάρχει και αυτό το εμπόδιο και θα πρέπει να, ξεπερα... να ξεπεραστεί. Είμαστε μια μεγάλη συμμαχία λοιπόν και αυτό πιστεύω ότι μας ενώνει, μας ενώνει και με τους εθνικούς βουλευτές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και χαίρομαι που την κάνουμε. Ανυπομονώ να ακούσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θέλω να βελτιωθούν λοιπόν οι σχέσεις μας, γιατί νομίζω ότι έτσι θα ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ενισχύσουμε και τη δημοκρατία στην Ευρώπη με το σχηματισμό αυτών των συνασπισμών της Συμμαχίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, πρέπει να φύγω για λίγο. Παρακαλώ τον Σέλφο Μέσοστε να, να, πάρει το λόγο, να πάρει την ε, θέση μου στην Προεδρία και η κυρία Τέιν έχει το λόγο. ο κύριος Νταφ μάλλον. Όχι. Ναι, ναι, έχετε, έχετε δίκιο κυρία Τάιν, εσείς έχετε το λόγο. Κύριε Μαρτίνες, και εγώ να σας πω χρόνια πολλά εκ των υστέρων και κυρίως να σας ευχαριστήσω για το ανοιχτό πνεύμα και για την επικόνηση της κατάστασης που είναι πολύ σημαντική θεωρώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, πρόταση του Δανεικού Κοινοβουλίου να χρησιμοποιούμε μόνο δύο γλώσσε. Νομίζω ότι υπάρχεται στην γενικότερη απόπειρα εξοικονόμηση κόστου και σίγουρα πρόκειται για ένα από τα θέματα τα οποία και έτσι ε, συμβάλλουν στο χάος που δημιουργείται και στη Γερμανία. Για παράδειγμα, για την πολυγλωσία, για την διπλή έδρα, όλα αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε την εξοικονόμηση του κόστους, γιατί θεωρώ ότι η αύξηση του προϋπολογισμού και τα ποσοστά που έχουμε, δεδομένου και του γεγονότος ότι γίνονται ε, μέτρα λιτότητα και γίνονται μέτρα έτσι εξοικονόμησης από όλες τις κυβερνήσει. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν να κατανοήσουν λοιπόν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Για να περάσω όμω στο θέμα που μα απασχολεί Νομίζω ότι η τάση επαναθνικοποίησης δεν μπορούμε να την αρνηθούμε και σε ό,τι αφορά την αρχή της επικουρικότητας. Μια υπουργό στη Γερμανία είπε ας αφήσουμε και λίγη δουλειά στους, Ευρωπαίους, ε, στους, Ευρωπαϊκούς, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια τάση η οποία θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με το ότι μας θεωρούν αντιπάλους. Όχι, δεν είναι θέμα ε, παιχνιδιού εξουσίας. Όχι, μιλάμε και για φόβο, γιατί έχουμε την ευρωπαϊκή κρίση, την ε, οικονομική κρίση. Και να σας πω ότι για τη δική μου χώρα τουλάχιστον αυτό προκαλεί φόβο στον κόσμο. Γιατί πολλοί κόσμοι θεωρούν ότι προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει να το λάβουμε σε σοβαρά τους φόβους αυτούς. Ιδιαίτερα επειδή ω τώρα δεν το έχουμε καταφέρει ως Ευρωπαίοι βουλευτές ε, σε εθνικό επίπεδο και στα εθνικά μέσα να προβάλλουμε τη δουλειά μας επαρκώς. όπως οι εθνικοί βουλευτές. Και φυσικά είναι εξαιρετικά σημαντικές οι επαφές σε διμερές επίπεδο, όπως αναφέρθηκε σε όλα τα επίπεδα και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνονται ταξίδια συνέχεια προς όλες τις πρωτεύουσες, προς 27 πρωτεύουσες από πλευράς ε, των Ευρωπαϊκών Επιτροπών, αλλά ο Επιτροπός ΡΕΝ ε, ε, πήγε και μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι ήταν ο πρώτος επίτροπος ο οποίος παρευρέθηκε στο Ευρωπαϊκό Bundestag μετά από πέντε χρόνια. Πέρα από όσα είπε, βοήθησε στο να ξεδιαλυθούν διάφορες παρανοήσεις και γενικά έγινε πάρα πολύ θετικά δεκτή και η επίσκεψη του. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να το επιδιώξουμε αυτό σε ό,τι αφορά και θέματα τα οποία ε, προκαλούν ιδιαίτερο φόβο. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, σε ό,τι αφορά θέματα οικονομικής κρίσης, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό και ωφέλιμο. And then the last on the list, Mr. στον κατάλογο, ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ πολύ και πρέπει να ζητήσω γνώμη από τον ε, Μιγέλ Μαρτίνες ε, γιατί δυστυχώς δεν ήμουν ε, παρόν στην αρχή της συνεδρίασης αλλά έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά, κατανοώ πλήρως τη θέση, και, τη θέση του και την συμμερίζομαι. Όμως θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλες τις υποεπιτροπές οι οποίες ήρθαν στο Westminster την Πέμπτη Ελπίζω ότι δεν ε, ήταν ιδιαίτερα τραυματική ή μάλλον όχι δεν ήταν υπερβολικά τραυματική η εμπειρία. Αλλά βεβαίως η μέρα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, και κατέστη σαφές το χάσμα που υπάρχει μεταξύ μας ανάμεσα στο Westminster και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, είναι σαν ε, να έχουμε δύο διαφορετικές τροχιές οι οποίες μπορεί κάποια στιγμή ε, να ταυτιστούν αλλά όχι προγραμματισμένα, μάλλον τυχαία. Εν πάση περιπτώσει μπορώ να πω ότι σε όλες τις πολιτικές ομάδες μεγαλώνει η απόκληση ανάμεσα στην ε, πολιτική τάξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας το θέσω έτσι, και τους εθνικούς βουλευτές. Και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε, τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να το θέσω σαν κεντρικό ζήτημα στην ε, πολιτική ε, συζήτηση που κάνουμε. οι εξελίξεις ε, στα εθνικά, στις εθνικές δομές δεν καταλαβαίνουν μερικές φορές, δεν κατανοούν ότι μπορεί να επηρεάσουν το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Και στη Βουδαπέστη κάποιες ε, αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της ε, Γερμανίας ε, μπορούν να βρουν υποστηριχτές ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ξέρετε ότι από τη στιγμή που ξεκινά η διαδικασία ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία να περνάει από τον έλεγχο του, ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό θα γίνεται συστηματικά στο Westminster και ενδεχομένω ε, συστηματικά θα μπλοκάρονται κάποιες ε, αποφάσεις. Και είναι γεγονός ότι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους έτσι ώστε να ξεπεραστεί το βρετανικό βέτο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ στην Επιτροπή μας. Δηλαδή να δούμε πολύ προσεκτικά το ενδεχόμενο ε, αντίδρασης στην ε, αγγλική απόφαση, στην βρετανική απόφαση να αλλάξει η διαδικασία έγκρισης όλων των εξελίξεων που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Βεβαίως είναι ορθή και η πρόταση που έγινε, έστω και αν είναι χρονοβόρα, να επισκεπτόμαστε τις διάφορες πρωτεύουσες, να ερχόμαστε σε επαφή με τα κοινοβούλια. Φυσικά πρέπει να μιλάμε ε, και σε, σε φόρα τύπου Κόζακ, αλλά πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή και με τα εθνικά κοινοβούλια μετακινούμενοι προς αυτά, δηλαδή να πηγαίνουμε στις χώρες τους. Νομίζω ότι η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τη δομή της Λισαβόνας είναι οι διαπραγματεύσεις για την μεταρρύθμιση του προπολογισμού. Η τροποποίηση δηλαδή των πολιετών δημοσιονομικών ε, προοπτικών και η τροποποίηση του συστήματος ε, ιδίων πόρων. Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία πρόοδο στα θέματα αυτά, εάν υπάρξει απλώς αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ιδίως σε μια χρονική στιγμή όπου Uh, όπου η θέση της Επιτροπής είναι μάλλον ε, ευκαιριακή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δουλέψουμε λίγο την ιδέα ε, μιας διάσκεψης ε, που θα αφορά τα δημοσιονομικά, τον προϋπολογισμό, τις δημοσιονομικές προοπτικές και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια διάσκεψη ε, σύμφωνα και με τις προτάσεις εκθέσεως Γκουελπιέρη υπό το 2.36. Τέλος, πιστεύω ότι η Βελγική Προεδρία πλήρως κάλυψε τη θέση της, δηλαδή ε, καλής συνεργασίας για θέματα ΚΕΠΑ. Και ελπίζω ότι τουλάχιστον από εκεί κάτι επικοδομητικό θα προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντάφλε, ο Πρόεδρος. Στην ε, επόμενη συνεδρίαση θα μας πείτε πώς έγινε η, πώς, πώς προχώρησε η συνάντηση των μαθηματικών όλου του κόσμου στο Κέμπριτζ. Τώρα θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Εγώ δεν ήμουν στο Κέμπριτζ, αλλά δεν έχει σημασία. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες για να απαντήσει στα διάφορα ερωτήματα τα οποία προέκυψαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να πω πάντως και να τονίσω το ενδιαφέρον της συνεδρίασης αυτής. Να πω ότι Ποτέ δεν είχα ξαναέρθει στην επιτροπή σας, φίλε Καζίνη, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και με ικανοποίησε ιδιαίτερα και το επίπεδο ε, της σακφήνειας, της ακρίβειας, οι απόψει συναδέλφων που προέρχονται από τελείω διαφορετικές ε, πολιτικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα επίπεδο ομοιογένειας πάρα πολύ αξιοσημείωτο τουλάχιστον σε σχέση με αυτό το οποίο εγώ περίμενα. Ένα από τα πράγματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρα μετά από τις παρεμβάσεις πολλών από τους ε, συναδέλφους είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κόζα συγκεκριμένα και γενικότερα στις σχέσεις μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ουσιαστικά η κορυφή του παγόβουνου. Ένα σύμπτωμα, αν θέλετε, μιας κατάστασης όπου φαίνεται να υπάρχει μια αποσύνθεση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, θα ήταν καλύτερα έτσι, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε κάποιος να παρέμβει και να επιλύσει πολύ πιο εύκολα το θέμα. Όχι. Έχετε δίκιο λοιπόν. Είναι η προβολή ενός προβλήματος ή μια σειράς προβλημάτων πολύ σοβαρότερων τα οποία αντιλαμβάνεστε από ό,τι φαίνεται εδώ εσείς όλοι ή περισσότερο από εσάς. Και πράγματι είναι σοβαρή η κατάσταση, είναι σοβαρά τα προβλήματα. Ο κύριος Γκερέρο μας μίλησε για τα διάφορα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται και τα οποία δυσχεραίνουν αυτού του είδους της διασυνδέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Και φυσικά συμφωνώ, συμφωνώ ιδιαίτερα με όλες αυτές τις δυσκολίες που αναφέρατε κύριε Γκερέρο. Όλες όμως αυτές οι δυσκολίες πρέπει να πω ότι ουσιαστικά ε, επιδεινώνονται και σε αυτό το γενικότερο κλίμα που είναι ε, η απώλεια αν θέλετε ελπίδας και επίστης σε αυτή τη διαδικασία της δυτικής οργάνωσης που για κάποιους είναι απλά απολύτως αναγκαίο για να ιδρυωθεί και η πρόοδος σε καθέναν από τους λαούς μας. Μπορεί κανείς να είναι φιλοευρωπαϊστής γιατί έχει κάποια ιδεολογική τέτοια τοποθέτηση. Ε, δεν είναι στο αίμα μας αν θέλετε, δεν είναι κάποιος γενετικός λόγος. Ο βασικός λόγος είναι ότι είμαστε πεπισμένοι ότι η πρόοδος του λαού μας σε καμιά περίπτωση στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης και των πολυμερών σχέσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εδρεωθεί εάν η χώρα μας δεν μπορεί μέσα σε μια πολύ πιο σε μια ζώνη πολύ μεγαλύτερης επιρροής μπορεί να δράσει μόνη Φυσικά δεν μπορεί να δράσει μόνη της η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Γερμανία ακόμη περισσότερο. Δεν μπορούμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών απομονωμένοι ο καθένας. Έχουμε και θέματα σταθερότητας και οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν μπορούν αυτά να ευρώθουν σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, εκεί πιστεύω ότι υπάρχει ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον από τους ευρωσυμπατριώτες μου, εκτός αν δεν πιστεύουν στο σχέδιο στο οποίο πιστεύω εγώ, οι οποίοι πιστεύουν ότι αν συμμετέχουν μόνοι τους στο σκέλος που αντιπροσωπεί η δική τους χώρα, η περιοχή, η περιφέρεια, θα μπορέσουν αυτόν τον τρόπο μόνοι τους, να προασπίσουν τα συμφέροντα και την πρόοδο των πολιτών της χώρας τους. Δεν μπορώ πώς χωράει στο κεφάλι κάποιου βλέποντας ε, τον κόσμο, βλέποντας που είναι η Κίνα σήμερα, που είναι η Βραζιλία, που είναι η ΙΠΑ, να πιστεύει ότι μόνος του ε, ας πούμε το Λουξεμβούργο, για να αναφέρω μία μόνο χώρα, ότι μπορεί να προχωρήσει και να επιτύχει τη γενική πρόοδο, την πρόοδο όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Λοιπόν, βγαίνοντα από αυτή την εντύπωση που νομίζω την επιβεβαιώνετε και όλοι εσείς ότι δηλαδή εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα συγκεκριμένο αλλά με σύμπτωμα μία σειράς προβλημάτων ε, ή τέλος πάντων με πολύ πιο βαθιά και ουσιώδη προβλήματα υπάρχει κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή φαίνεται να τονίσατε όλοι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μία τεράστια έλλειψη και αδυναμία σε αυτό το οποίο εμείς κάνουμε. Και τι αντιλαμβάνεται και η κοινή γνώμη σε σχέση με αυτά που κάνουμε. Δηλαδή, από ό,τι κάνουμε εμείς εδώ, ούτε κάνουν στους συμπατριώτες μας, τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, δεν φτάνει αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν φτάνει εκεί. Δεν φτάνει ούτε στους συντρόφους μας από τα εθνικά κόμματα. Πάρα πολύ καλά τα είπατε κύριε Νταφ αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα είναι ότι οι βουλευτές της χώρας μας, της ίδιας χώρας, του ίδιου πολιτικού κόμματος, στο οποίο ανήκουμε εμείς από το εθνικό επίπεδο όμως, δεν γνωρίζουν εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Τι κάνουμε εμείς οι ευρωβουλευτές που προερχόμαστε από την ίδια χώρα με αυτούς και από το ίδιο πολιτικό κόμμα με αυτούς. Δεν το γνωρίζουν. Αν δεν το γνωρίζουν πώς θα το εκτιμήσουν, πώς θα το αξιολογήσουν. Ακούστε πράγματι, αυτό είναι ένα θέμα που εμείς πρέπει να το λέμε εδώ, γιατί υπάρχει και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και μία από τις λύσεις, ή τέλο πάντων από τις συνταγές για την αντιμετώπιση του προβλήματος, είναι να το δούμε και στις δικές μας πολιτικές οικογένειες, ή ορισμένες από τις πολιτικές οικογένειες. Από εκεί περνάει η λύση του προβλήματος. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ομάδα ε, στην οποία ανήκω πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το ίδιο πρέπει να κάνει το ΕΛΚ, το ίδιο πρέπει να κάνουν οι πράσινοι. Πρέπει δηλαδή να μπορέσουμε να είμαστε ικανοί να καθιερώσουμε κάποιου μηχανισμού, ε, επαρκεί μηχανισμού επικοινωνία μεταξύ μα ώστε τουλάχιστον οι δικοί μα ε, σύντροφοι από την ίδια πολιτική οικογένεια και από την ίδια χώρα να γνωρίζουν τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει εδώ στην Ευρώπη. Και εκεί υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά δαπανά πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα για την επικοινωνία και νομίζω ότι αυτή η άσκηση και αυτό το εγχείρημα δεν είναι καθόλου αποδοτικό. Έχουμε όλο και περισσότερα μέσα, όλο και περισσότερες τεχνολογίες, όλο και περισσότερους μηχανισμούς. Όχι όμως μεγαλύτερη γνώση, μεγαλύτερη εκτίμηση ή μεγαλύτερη και καλύτερη επικοινωνία με τους ε, συμπολίτε μας. Και νομίζω το είπε ο κύριος Σόντεργαρτ. Δεν γνωρίζουν όχι μόνο τι γίνεται στο κοινοβούλιο, αλλά και το τι γίνεται γενικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ε, φαντάζομαι ότι ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποιο λάθος έχει γίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γιατί μιλάω. Μιλάω για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια ήταν ένα ασφάλμα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερόπτε και αλαζονικοί. Ε, ίσως ε, προβάλαμε τους πόρου που έχουμε, ότι είναι πάρα πολλοί πόροι και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή μα. Κάποιο λάθος κάναμε, γιατί πραγματικά δεν δικαιολογείται διαφορετικά αυτή, ε, αυτός ο φόνος που είδα και τον οποίο δεν είχα συνειδητοποιήσει αρκετά τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ πάρα πολύ καλά τα είπε και μετρημένα ως συνήθως. Ε, είπατε εσείς ότι διαφωνούμε. Όχι, εγώ νομίζω ότι συμφωνούμε. Πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να έχουμε διάλογο και βέβαια να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς προκαταλήψεις. Τέλο πάντων με τις ελάχιστες δυνατές προκαταλήψεις. Είμαστε δημοκράτες. Φυσικά και είμαστε πεπισμένοι ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία. Αυτό που πιστεύω όμω είναι ότι σε ό,τι αφορά τη μορφή, σε ό,τι αφορά τη μορφή διάρθρωσης αυτή της συνεργασίας για την οποία μας υποχρεώνει η συνθήκη, η φόρμουλα που πρότεινα εγώ είναι πρώτα απ' όλα να αφήσουμε την ΚΟΣΑΚ ως έχει, ε, όπως λειτουργεί, να εργαστούμε, να εξορθολογήσουμε, αλλά σας είπα κατά δεύτερον ότι για συγκεκριμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα οποία αναφέρθηκε ο Άντριου Νταφ, και θέματα πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, εκεί νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ δύο εναλλακτικών. Η μία είναι, όπως είπα πριν, να δούμε πώς μπορούμε να ταιριάξουμε, να βάλουμε έναν μηχανισμό που δεν μπορεί να είναι ένας από τη μία πλευρά, 40 από την άλλη, πρέπει να είναι ένας καινούριο, πιο ισορροπημένος μηχανισμός. Ή άλλη αναλλακτική που μπορούμε να επιλέξουμε και η οποία ειλικρινά σας το λέω μου φαίνεται λογική, είναι η εξή να πούμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια συμφωνούν μεταξύ τους και καθιερώνουν το μηχανισμό τον οποίο θέλουν για τις συζητήσεις τους, για το διάλογο, για τη λήψη αποφάσεων και όταν αυτοί θα έχουν λάβει τις αποφάσεις τους και όπως και εμείς από τη δική μας πλευρά θα κάνουμε τις δικές μας συναντήσεις και θα, θα αποφαινόμαστε από μόνοι μας, μετά θα συναντιόμαστε και οι δύο αλλά με ισομερή εκπροσώπηση και με καλή πρόθεση, με ανοιχτό πνεύμα, σε όσμωση, αν θέλετε, να συζητούμε. Αλλά δεν δέχομαι για αυτή τη συζήτηση μια δομή όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει να αντιμετωπίσει 40 διαφορετικά οράματα που κάθε ένα από τα οποία εκπροσωπεί αυτό που μπορεί να εκπροσωπεί. Φυσικά και δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός, φυσικά και δεν πρέπει να υπάρχει λογοκρισία στα θέματα τα οποία συζητούμε ή στο πνεύμα συζήτησης. Ο κύριο Σόντεγκαρτ νομίζω ότι πολύ ε, ξεκάθαρα επισήμανε την αποτυχία και στην επικοινωνία αλλά και στην εκπαίδευση. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Είναι προφανές ότι κανένας από τους οργανισμούς και από τις οργανώσεις, από τις κοινωνικές οργανώσεις. Ε, καμία οργάνωση δεν προωθεί έτσι μια φιλοευρωπαϊκή εκπαίδευση και παιδεία. Και δεν είναι πρόσφορο το έδαφος αυτό για να προχωρήσουμε. Και έχετε και βέβαια δίκιο όταν λέτε ότι φυσικά η αντίσταση που συναντάμε, που μπορεί να συναντήσουμε, γιατί διάφοροι αποφασίζουν και παρεμβαίνουν σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα που ο κύριε Σόντεγκαρτ θα το έθετα λίγο διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει αποφάσει που επηρεάζουν τι χώρε μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσει. Τι αποφάσει τι λαμβάνει το Συμβούλιο ή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με του νέου τόμει απόφαση που έχουμε. Δεν είναι η Κομισιόν αυτή η οποία ούτε επιβάλλει στη, που δεν επιβάλλεται στην Ισπανία, στην Δανία. Πολύ εύκολα μπορεί κανεί να το πει αυτό, γιατί και εγώ το έχω ακούσει στην Ισπανία. Όχι, δεν το κάνουμε εμεί. Η Βρυξέλλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει. Όχι. Πρέπει να πάρουμε τι ευθύνε μα κι εμεί. Ή το Συμβούλιο ή Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θεσπίζουν αυτά τα οποία θα επηρεάσουν μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Ισπανία κτλ. Ο κύριος Ρανζέλ δεν είναι στην αίθουσα πια, αλλά πάντα όσα λέει είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και ανέφερε και κάτι σχετικά με την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των, Ευρω... των Εθνικών Κοινοβούλων, κάτι που θίξατε και αρκετοί άλλοι από εσάς. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι η ανομοιογένεια μεταξύ των διαφόρων Εθνικών Κοινοβουλίων έχει ως αποτέλεσμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεθνικά κοινοβούλια συνολικά και στο επίπεδο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με καθένα ξεχωριστά από τα εθνικά κοινοβούλια, έχουμε δυσκολίε. Γιατί ακριβώ αυτή η ανομοιογένεια που υπάρχει. Πώ να το εκφράσω. Έχουμε το Ιταλικό Κοινοβούλιο όπως έχει εκλεγεί και τα λοιπά. Έχουμε τη Βουλή των Λόρδων από την άλλη πλευρά που δεν εξέλεξε κανείς τα μέλη της. και δεν έχει και πολλές αρμοδιότητες ε, στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα ασχολείται πολύ περισσότερο με τα ευρωπαϊκά θέματα. Να μην μιλήσουμε για τώρα για διαφορά μεταξύ Μπούντεστα και Στονικού ή Δανικού Κοινοβουλίου, αλλά ε, εννοώ το εξή. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δυσκολεύεται ή θα δυσκολευόταν να συστήσει έναν μόνιμο μηχανισμό διαμεσολάβησης και διάδραση με όλα τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά υπάρχουν και μία σειρά εθνικών κοινοβουλίων που δεν έχουν καμία δυνατότητα και καμία ικανότητα για τη θέση αυτή μόνιμη επικοινωνία ε, σε καθένα από τα θέματα. Το δικό μου κοινοβούλιο ε, είναι ένα από τα μεσαία προς μεγάλα κοινοβούλια. Και δεν μπορεί συνέχεια παρόλα αυτά να είναι σε συνεχή διάδραση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το φαινόμενο ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Κύριος ε, Σέπλιν, πάντοτε μετρημένος, ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τα σχολιά του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει αρκετή γνώση για αυτά που κάνουμε. Λείπει αυτή η γνώση. Αλλά μπορεί να αποκτηθεί γνώση αυτή πρώτα. Όταν εμείς από μόνοι μας πάρουμε στα σοβαρά την ανάγκη επικοινωνία και αρχίσουμε να επικοινωνούμε και αν βέβαια πετύχουμε από την άλλη πλευρά και τα μέσα επικοινωνία να ενδιαφερθούν πραγματικά για αυτά που κάνουμε. Ακούστε, εγώ υπήρξα μάρτυρας, βίωσα ε, στο κοινοβούλιο μια στιγμή όπου μια συνάδελφός μας με το που σηκώθηκε για να πάρει το λόγο ε, πιάστηκε η φούστα της ε, στο έδρανο και βρέθηκε με το εσώρουχο στη μέση, μπροστά στο να μιλήσουν προς στον κόσμο. Και τα μέσα επικοινωνίας τότε έδωσαν μεγάλη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί βρέθηκε μία συνάδελφος με το εσώρουχο μπροστά στο μικρόφωνο. Εντάξει, μπορούμε να γελάσουμε, αλλά είναι λυπηρό, είναι θλιβερό γιατί υπάρχουν εδώ ανταποκριτέ από όλα τα μέσα επικοινωνίας Και ποιο ήταν το θέμα που ενδιέφερε πιο πολύ την κοινή γνώμη της χώρας μα, αυτό που σα είπα. Είναι λίγο γκροτέσκο, θα το πω. Ε, είναι λίγο γελίο γιατί αυτά είναι τα μέσα επικοινωνίας με τα οποία εμείς δουλεύουμε κάθε μέρα του χρόνου. Είναι ανησυχητικό. Και τι πρέπει να κάνουμε, να σοπάσουμε, φυσικά και όχι, το αντίθετο, πρέπει να εργαστούμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και εμένα θα με ανησυχούσε εάν δεν έρχονταν ε, συνάδελφοι και από τα παλιά κοινοβούλια και έρχονταν μόνο από τα ε, καινούρια. Άκουγα ε, τους παλιούς αλλά άκουσα και τον ε, συνάδελφο από την Ουγγαρία που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Έχουμε και τα προβλήματά μας με την Ουγγαρία αλλά είναι τα ίδια με αυτά που έχουμε και με την Ισπανία και με τη Γερμανία. Στις σχέσεις μας εννοώ. Και αυτά που μας είπε και ο κύριος Γκρότ είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως πάντοτε άλλωστε. Και πρέπει να πω ότι οι πολιτικές ομάδες σίγουρα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που δεν έχουν αναλάβει μέχρι στιγμής. Κανένα από τα κόμματά μας. Και εμένα με ενδιαφέρει πολύ γιατί η Γερμανία έχει ε, δυνατότητες και δυναμικό ώστε να, είναι, ε, να χρησιμεύει ως υπόδειγμα για όλους μας. Για το πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα σε χώρες που έχουν παράδοση κοινοβουλευτική μακρόχρονη σε χώρες που πρωταγωνίστησαν ε, σε όλη τη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Τι κάνετε εσείς δηλαδή για να γίνει πραγματικά γνωστό καθημερινά το ευρωπαϊκό φαινόμενο, όχι μόνο στην κοινή γνώμη, αλλά και στους εθνικούς κοινοβουλευτικούς ε, και περιφερειακούς ε, φορείς. Ίσως είναι λίγο τολμηρό αυτό, ίσως θα πρέπει να το πω στο Προεδρείο, ότι ίσως πρέπει να ξανατεθούν τα προγράμματα που έχουμε με τις ομάδες επισκεπτών, να τα ξανασυζητήσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα για ομάδες ε, επισκεπτών που περιορίζονται στο να κάνουν ε, έτσι επισκέψεις, να δουν πώς είναι η αίθουσα αυτή, πώς είναι το κοινοβούλιο, πώς είναι η ολομέλεια, αλλά δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε ή όσο θα μπορούσαν αυτές οι επισκέψεις ώστε πραγματικά ο στόχος να είναι αυτοί που έρχονται να είναι άτομα τα οποία πραγματικά θα μπορούσαν στη συνέχεια να επηρεάσουν. Και όχι να φέρνουμε κάποιους ή κάποιους νέους, κάποιους φοιτητές, ε, έτσι σαν βραβείο. Και να μην το πρόγραμμα δύο ή τρεις ώρες μόνο, αλλά πραγματικά μία μέρα ολόκληρη και να βλέπουν πραγματικά οι επισκέπτες μας τι γίνεται, πώς γίνεται και βέβαια να ε, μπορούν μετά να τα ε, μεταφέρουν. Για την κυρία Τέι, Να σας πω καταρχάς ότι στο έργο το οποίο κάνουμε εδώ πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε και την καταπληκτική δουλειά της κυρίας Σιλβάνα Κόρχ Μερίν που πραγματικά κάνει καταπληκτική δουλειά. Είναι από τη χώρα σας, ε, είναι συμπατριώτησά σας, κάνει καταπληκτική δουλειά. Ε, θέλω να σας πω σε σχέση με τις γλώσσες. Είμαι σίγουρος ότι κανένας από τους συναδέλφους βουλευτές αλλά και κανένας από τους εδώ παρόντες δεν μπορεί να μας πει πόσο κοστίζει η πολυγλωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Γιατί γίνεται πολλή λόγο. Πόσο κοστίζει όμω, Πόσο κοστίζει κάθε, για κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να διαβάζει όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γλώσσα του. Πόσο κοστίζει κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει εκπροσώπους δεν είμαστε στο μπάσκετ να διαλέγουμε αυτούς που είναι πάνω από δύο μέτρα. Εδώ οι βουλευτέ δεν τους επιλέγει, δεν τους ψηφίζει ο κόσμος γιατί μιλάνε δύο ή τρεις γλώσσες, αλλά γιατί αξίζουν την εμπιστοσύνη των συμπολιτών τους για να τους εκπροσωπήσουν εδώ και να προασπίσουν τα συμφέροντά του εδώ. Και μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην ξέρουν παρά μόνο τη μητρική του γλώσσα. Όλες οι δαπάνε για διερμηνία και μετάφραση σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοστίζουν ένα καφέ, ένα φθηνό καφέ για κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σας παρακαλώ να το πείτε αυτό. Ο ένας καφές φθηνός, ένα ευρώ μιλάμε τώρα έτσι, για ένα ευρώ. Θα μου πείτε βέβαια πού κοστίζει ένα καφέ σε ένα ευρώ. Και στη χώρα μου θα ψάξω πολύ για να το βρω. Αλλά τέλο πάντων, τόσο κοστίζει η τιμή ενό καφέ. Τόσο κοστίζει η διερμηνία και στι 23 επίσημε γλώσσε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο Κοινοβούλιο. Ένα ευρώ ανά Ευρωπαίο πολίτη και ανά έτος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πάρα πολύ φθηνό. Φυσικά, όταν κάποια στοιχεία τα παρουσιάζουμε έτσι απομονωμένα και λέμε ότι είναι 500-650 ε, εκατομμύρια ευρώ, ε, είναι πολύ όταν το ακούμε έτσι, αλλά σε πραγματικό αριθμό, πραγματικά, σε πραγματικούς αριθμούς είναι η τιμή ενός καφέ, ενός φθηνού καφέ, κατά κεφαλή και αναέτος. Και αυτή είναι η τιμή που πληρώνουμε για τη δημοκρατία. Εσείς μπορεί να πείτε πολύ ωραία αγγλικά αλλά μπορείτε να μας τα πείτε στη γλώσσα σας και μπορούν να σας ακούσουν και τα εκατομμύρια Γερμανοί συμπολίτε σας στη γλώσσα σας για να καταλάβουν τι λέτε. Αν σας ακούσουν αγγλικά, λίγοι θα σας καταλάβουν, πολλοί δεν θα σας καταλάβουν. Και υποθέτω ότι μιλάτε και τέλεια αγγλικά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα θέμα τόσο σημαντικό από ιδεολογικής πλευρά σε σχέση με τις αρχές που διέπουν, που μας διέπουν θέλεις, αυτή τη διαδικασία που πραγματικά με τα λόγου γνώσεως και με πολύ μεγάλη μετριοπάθεια πρέπει να τα συζητήσουμε γιατί πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε τελικά. Κάνατε και ένα τελευταίο σχόλιο το οποίο μου φαίνεται εμένα προσωπικά ιδιαίτερα σημαντικό και το σημειώνω. Το σημειώνω γιατί ίσως δεν ήταν ξεκάθαρο για μένα. Δηλαδή, σημασία, τη σημασία που έχει ε, Είπατε για επιτρόπους, μπορεί να θέλατε να εννοήσετε κάποιους άλλους ανώτερους αξιωματούχους που λέτε ότι τι σημασία έχει που πηγαίνουν στα Εθνικά Κοινοβούλια ή επίτροποι και μιλάνε. Είναι ενδιαφέρον στοιχείο αυτό, πρέπει να το σημειώσουμε. Και κοιτάξτε, η ανησυχία μου είναι η εξή. Είναι το ίδιο. Ένα επίτροπο, αν πηγαίνει στην Bundestag, και με εξέπηξε λίγο αυτό που είπατε εσεί, ε, ότι σε πέντε χρόνια ένας επίτροπος πήγε και είχε επαφές με τους ε, Γερμανούς βουλευτές. Φυσικά και με κλείσει αυτό θα έπρεπε να πάει πολύ συχνότερα. Αλλά θα με εξέπλητε επίσης ένας επιτροπός να πηγαίνει να μιλάει στο Εθνικό ε, Κοινοβούλιο και αντί να συναντά 50 βουλευτές, να συναντά 4. Γιατί οι βουλευτές της εν λόγω χώρας έχουν τελικά 40 επίγοντα θέματα άμεσης σημασίας τα οποία πρέπει να τα συζητήσουν και δεν πηγαίνουν στις συναντήσεις με τον Επίτροπο. Όπως συμβαίνει και εδώ, είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε να τη συζητήσουμε μεταξύ μας. Αλλά όχι και να την μεταφέρουμε έτσι και πολύ προς τα έξω. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Νταφ, που με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο θα έλεγα, υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό και στο οποίο έκανε αναφορά και ο κύριος Νταφ. Είναι το θέμα της συζήτησης μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Είναι ένα καθοριστική σημασία ζήτημα και θα ήταν σκόπιμο χωρίς ε, φόβο και χωρίς ε, βιασύνη να το αναφέρουμε έτσι χαλαρά να το συζητήσουμε με όλα τα στοιχεία και με όλες τις επιλογές που μπορεί να τεθούν από εδώ και πέρα. Κύριε Ντάφ, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που όλοι μας θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Είναι μια θεμελιώδης πρωτοβουλία, πρέπει να την κοινοποιήσουμε και πρέπει να ε, την προωθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πρόεδρε, σε ευχαριστώ εσένα για την αξιοσημείωτη υπομονή σου. Έφυγε δυστυχώς ο φίλος Αρανιζέλ. Ε, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για την Παλαιά Διαθήκη, κάτι ανέφερε ο κύριο Ρανζέλ. Εγώ θα ήμουν πιο πολύ τη καινή διαθήκη, αλλά νομίζω ότι ε, έχεις και εσύ υπομονή, η όβιο. Είναι μάλλον ε, μια αρετή φλωρεντιανή Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε σήμερα να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας και βασίζομαι στους κυρίους Νταφ και Κουαλτιέρη για να δούμε τι θα πούμε για το ρόλο του εγγράφου αυτού του, το οποίο στέλνει και σε εμά αλλά και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια η Βελγική Προεδρία, το Βελγικό Κοινοβούλιο, για να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τη ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερικών και άμυνας και ασφάλειας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η συμμετοχή μου στην Επιτροπή σας. Εγώ ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες. Ευχαριστώ λοιπόν γιατί σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες ε, έδωσες και μία παθιασμένη γεύση. Είναι γεγονός ότι ε, εμείς πιστεύουμε σε αυτές τις βαθιές ρίζες που ε, αποτελούν τη βάση της Ευρώπης. Αυτές τις βαθιές ρίζες που φτάνουν, που φτάνουν στα ίδια τα σπλάχνα της Ευρώπης. Μοιραζόμαστε όλοι εδώ αυτό το ίδιο πάθος. Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετώ λοιπόν. Eh, λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα-δυο θεματάκια εμείς. Έχω και μια εκθεσούλα, λέει ο Πρόεδρος, για την ερμηνεία του άρθρου 51 του κανονισμού. Εγώ όμως σας προτείνω, μια και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να συζητήσουμε σήμερα το θέμα της τροποποίησης του κανονισμού που εγκρίναμε ε, σε σχέση με την πρωτοβολία των πολιτών. Ε, ναι, Πρόεδρε, για το θέμα αυτό η κυρία Γκουρμά, η οποία δεν είναι εδώ μαζί μας, γιατί έπρεπε να πάει σε μια επιτροπή. Επομένως, ε, μου ανέθεσε να σας παρουσιάσω το αίτημα της προς την Επιτροπή να εγκρίνουμε τη διόρθωση αυτή Πρόκειται για ένα τυπογραφικό λάθος ουσιαστικά σε σχέση με το κείμενο της πρωτοβουλίας, της νομοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών. Και αυτό το λάθος ουσιαστικά μας απομάκρυνε και από την πολιτική συμφωνία. Ποιο είναι το λάθος τώρα. Η αναθεώρηση μετά από τρία χρόνια της λειτουργίας αυτής της πρωτοβουλίας πρέπει να ξεκινά να μετράνε αυτά τα τρία χρόνια από την ημερομηνία εφαρμογής υποβολής αίτησης αυτής της πρωτοβουλίας ένα χρόνο μετά την ε, θέση σε, σε ισχύ. Ο κ. Πρόεδρος είχε υποβάλει την σχετική τροπολογία, είχε κάνει μια πρόταση δηλαδή πραγματική εφαρμογή να έχουμε αυτή την αναβολή 12 μηνών ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν τις ε, απαραίτητες αποφάσεις για την εφαρμογή της. Άρα η αναθεώρηση ξεκινάει, ουσιαστικά γίνεται μάλλον τέσσερα χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ και όχι τρία χρόνια μετά τη θέση ισχύς. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν στην Επιτροπή μας αυτή την απόφαση ώστε η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να λάβει μετά και αυτή την σχετική απόφαση και όταν το Συμβούλιο με τη σειρά του πλέον λάβει την απόφαση διόρθωσης 14 Φεβρουαρίου να εγκρίνουμε αυτή την τροποποίηση και έτσι οι συνεισηγητές ζητούν, κυρία Κουρμάη, ζητούν τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής μας με βάση τη διαδικασία που θεσπίζει το άρθρο 216 του κανονισμού. Ε, λοιπόν, για να είμαστε σαφείς. Στο πρόγραμμα που υπέβαλα στην αρχή της Ολομέλειας είχα πει ότι θα συζητήσουμε μέχρι και το σημείο 5 και ότι αύριο θα συζητούσαμε το ζήτημα το οποίο ε, παρουσίασε εσύ, συνάδελφε Γκερέρο. Τέλο πάντων, παρουσίασε το θέμα, μα είπε ότι συμφωνεί και η κυρία Γκουρμάη, μάλλον μα εξήγησε ποια είναι η γραμμή σκέψη τη κυρία ε, Γκουρμάη και επομένω μπορούμε να αποφασίσουμε επί του σημείου αυτού που είναι το σημείο 11 και μετά να επανέλθουμε στο σημείο 5. Πρόκειται για μία καθαρά τυπική τροποποίηση βάσει του άρθρου 216 ήταν ένα ας πούμε τυπογραφικό λάθος. Ε, ε, ζητούμε λοιπόν την συνένεση των συναδέλφων. Εάν κανείς δεν ζητήσει να πάρει το λόγο, ε, τότε θεωρείται ότι... Α, μάλλον όχι, να κάνουμε μια ψηφοφορία. Α, ο Νταφ θέλει το λόγο. Κύριε Νταφ, παρακαλώ. Νομίζω πρωτού ψηφίσουμε επί των τροπολογιών, ε, επί του κειμένου, θα πρέπει να δούμε το κείμενο με όλο το σεβασμό, γιατί μπορούμε να το συζητήσουμε στους συντονιστές αυτό το πρωί. Αλλά εγώ δεν έχω λάβει κείμενο και θα πρέπει να το δω. Ε, Στο σημείο 11 υπάρχει το κείμενο. Στο σημείο 11 του φακέλου σας υπάρχει το κείμενο στο οποίο αναφέρθηκε ο συνέλφος Γκορέρο. Α, ορίστε, τώρα έχω το κείμενο. Δώστε μου λίγο χρόνο να το διαβάσω. Αν θέλετε, λέει ο Πρόεδρος, μπορούμε να σταματήσουμε πέντε λεπτά, να διακόψουμε πέντε λεπτά. Αλλά πραγματικά σας λέω, είναι πολύ απλή η τροπολογία αυτή. Και διαβάζω το κείμενο οι λέξεις «Τρία χρόνια μετά από την έναρξη ισχύω του παρόντος κανονισμού θα αντικατασταθούν από τις λέξεις «Τρία χρόνια από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού». 14 Φεβρουαρίου γίνεται τελικό το κείμενο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τα τρία χρόνια, όχι από την έναρξη ισχύω του κανονισμού, αλλά από την ημερομηνία, ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού εάν δεν ε, έχετε πρόβλημα, νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τη διόρθωση. Πάρα πολύ ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στο σημείο 5 το οποίο αφορά ένα κανονιστικό ζήτημα επί του οποίου έχω οριστεί εισηγητής. Στην ουσία πρόκειται για το εξής. Όπως γνωρίζετε, το άρθρο 51 προβλέπει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις, η διάσκεψη των Προέδρων έχει την αρμοδιότητα να ε, θέση σε δύο επιτροπές που εργάζονται από κοινού ε, σε κάποιο θέμα, να τους αναθέσει λέγω, να εκπονήσουν έκθεση από κοινού. Όμως ε, η διατύπωση αυτή δεν ήταν πολύ σαφής ε, και επομένως και οι συνάδελφοι Λάινε και λένε ως πρόεδροι επιτροπών πρόεδροι νομικής επιτροπής και περιβάλλοντος αντίστοιχα ζήτησαν από την δική μας Επιτροπή να απαντήσουμε σε τρία ερωτήματα. Πρώτον, να καθορίσουμε κατά πόσον αυτή η ενιαία εργασία από δύο ή και περισσότερες επιτροπές σε βάση του άρθρου 51 θα πρέπει να αφορά μονάχα την τακτική νομοθετική διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης ή και της άλλης φάσης. Δεύτερο ερώτημα να αποφασίσουμε κατά πόσον αυτή η από εργασία προϋποθέτει ότι και αρμοδιότητες που έχει στην Ολομέλεια η κάθε Επιτροπή να προτείνει απόσυρση κειμένου κτλ. τα λοιπά, οποιασδήποτε αρμοδιότητες ή εξουσίες έχει, μπορούν και πρέπει να ασκούνται ε, από κοινού ή όχι. Τρίτο ερώτημα. εάν αυτή η κοινή εργασία θα επιμηκύνεται και στις ε, ακόλουθες ε, φάσεις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης και εκτελεσκές πράξεις. Ο συνάδελφος Λένε πρότεινε κάποια διαφορετική ε, ερμηνεία βάσει μιας επιστολής που θα αποτελούσε με βάση της ερμηνείας. Ο κύριος Λάινε πρότεινε μια τροποποίηση. Εγώ προτείνω μια τροποποίηση του κανονισμού έτσι ώστε το άρθρο 51 από κοινού με τα άρθρα 50 και 49 κατά την άποψή μου χρήζουν αυτής της ε, τροποποίησης. Στο άρθρο 51 ας πούμε αναφέρεται ότι όταν ε, ε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 49 και 50 και εάν η διάσκεψη των Προέδρων είναι πεπισμένη ότι το θέμα είναι μεγάλης σημασίας, τότε μπορεί να ανατεθεί από κοινού η έκθεση κλπ. κλπ. Στην πραγματικότητα όμως, στο παρόν κείμενο των άρθρων 49, 50, 51 δεν ε, είναι σαφής ε, η διαφορά. Επομένως πρέπει κάπως να, αποφασι... να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Στο άρθρο 49 ναι, μπορούν να αναφέρουν τα θέματα απο των οποίων ενδεχομένως έχουν δείξει ενδιαφέρον παραπάνω από μία επιτροπή ε, θέματα για τα οποία αρμόδια καθήλυνη είναι μία επιτροπή αλλά χρειάζεται ή ζητά ε, την γνωμοδότηση μια αλλη επιτροπη Αυτή είναι μια απλή κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μία κεντρική επιτροπή η οποία είναι αρμόδια καθήλη. Στο άρθρο 50 προβλέπονται δύο υποθέσεις. Είτε ότι, ότι μία νομοθετική πρόταση περιέχει ένα σκέλος το οποίο αφορά σε μία επιτροπή και ένα άλλο σκέλος που αφορά μια κεντρικη επιτροπη η οποια ειναι αρμοδια καθηλυνη στο αρθρο 50 προβλεπονται δυο υποθεσεις ειτε οτι οτι μια νομοθετικη προταση επιτροπή και εκεί είναι πιο σαφής ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων. Και σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζεται ότι η αρμόδια είναι μία επιτροπή, αλλά η άλλη επιτροπή έχει ε, διευρυμένες, διευρυμένες αρμοδιότητες. Και επομένως οι τροπολογίες οι οποίες θα υποβληθούν από τη μία επιτροπή μπορεί να μην γίνουν ε, αποδεκτές από την άλλη ή ότι εν πάση περιπτώσει μπορούν από κοινού να υποβληθούν τροπολογίες στην Ολομέλεια. Η πρόταση που κάνω εγώ είναι να γίνει διαφοροποίηση ανάμεσα στο άρθρο 50 και 51 λέγοντας ότι το άρθρο 51 αφορά τις περιπτώσεις για τις οποίες είναι απολύτως αδύνατο να ξεχωρίσουμε ποια επιτροπή είναι αρμόδια καθήλυν. Σε περιπτώσεις λοιπόν που δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεχωρίσουμε τις αρμοδιότητες ε, και εάν και η διάσκεψη των Προέδρων βεβαίω συμφωνήσει ότι πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Εκεί μπορούμε, έτσι μπορούμε να αλλάξουμε το 51 έτσι ώστε να γίνει πιο σαφές. Να πούμε λοιπόν ότι οι προϋποθέσεις είναι δύο. Το θέμα το οποίο αφορά ε, τις αρμοδιότητες περισσότερων από μία επιτροπών και δεύτερον η διάσκεψη των Προέδρων να αποφανθεί ότι το θέμα ε, είναι μεγάλης σημασίας. Λοιπόν, από κοινού αρμοδιότητα δύο επιτροπών όταν και εφόσον είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τις αρμοδιότητες ε, των ε, επιτροπών με αυτήν την έννοια ε, δύο ή ενδεχομένως σε μια έκτακτη περίπτωση και παραπάνω από δύο επιτροπές ε, ξεκινούν μια κοινή νομοθετική διαδικασία. και κατά κανόνα ολοκληρώνεται με την πρώτη ανάγνωση αυτή η κοινή διαδικασία. Πάντως εάν ε, πρέπει να περάσει και σε επόμενη φάση σε κάποιες εξαιρετικές ε, περιπτώσεις όπου θα πρέπει να βρεθεί συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε συνεχίζει η κοινή διεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Όμως θεωρώ ότι όσον αφορά την τρίτη ερώτηση, δηλαδή ε, της κατα κατεξουσιοδότηση πράξης και τις εκτελεστικές, τότε από τη στιγμή που θα έχει συζητηθεί το θέμα, ε, μπορούν να απλωστευτούν οι διαδικασίες και επομένως είτε με αίτημα και των δύο επιτροπών είτε μετά από αίτημα ε, μίας από τις δύο επιτροπές ή ακόμα και από απόφαση ε, της διάσκεψης των προέδρων μονάχα μία επιτροπή να είναι υπεύθυνη για τις πράξεις αυτές. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ ως και όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόταση αυτή που μας υποβάλλατε. Κατά το παρελθόν Είχα και εγώ αντιμετωπίσει πολλέ φορέ το ζήτημα τη σύγκρουση ε, αρμοδιοτήτων μεταξύ επιτροπών και είχα υπάρξει θύμα. Επιτροπή Περιβάλλοντο, Επιτροπή Ιστορική Αγορά κτλ. Κανεί δεν ήξερε ποια επιτροπή θα είναι καθήλυνα αρμόδια. Και ίσω θα έπρεπε να προσθέσουμε και τη χρονική συνιστόσα, διότι κάποιε φορέ στο Συμβούλιο ήμασταν, ήταν πολύ πιο μπροστά, ενώ εμεί ακόμη στο Κοινοβούλιο ασχολούμαστε με το ποιο θα είναι αρμόδιο. Σω πρέπει να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα οι πρόεδροι των επιτροπών δεν μπορούν να συμφωνήσουν, θα μπορούμε να θετήσουμε την τάδε ή τη δίνα διαδικασία. Τώρα, δεν έχω να σας υποβάλω κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Ξέρω όμως ότι οι πρώτη των επιτροπών ε, ε ήταν, ε, είχαν πολύ δύσκολη δουλειά και σε ό,τι φορά την ενισχυμένη συνεργασία τι θα, ποιο θα είναι το αίτημα, τι θα υποβληθεί στην Ολομέλεια. Ήταν μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να υπάρχει κάποιο, κάποια χρονική προθεσμία προκειμένου οι διαδικασίες εδώ στο Κοινοβούλιο να περιορίζονται κάπως χρονικά. Το 1988 quando στο 188 μιλάμε για τα προτερήματα, μάλλον για την κατανομή των, των αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να εξετάσουμε αν είναι σωστή η κατανομή αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχει κανείς άλλος ερώτηση, νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε ε, την ε, προθεσμία για τις τροπολογίες. Α, κυρία Τάιμε, θέλει το λόγο. Ναι, θα ήθελα απλά να υποστηρίξω αυτά που είπε ο συνάδελφος, να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν ε, μεταξύ της Επιτροπής Καταναλωτών και Νομικών Υποθέσεων ε, διαμάχες για τις αρμοδιότητες και δεν προκύπτουν τα πράγματα αυτά χωρίς ε, συζήτηση και στην Επιτροπή Οίκων έχουμε προβλήματα γιατί είναι υπεύθυνη και αρμόδια για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει αντικείμενο θέματα που άπτονται των χρηματοπιστωτικών υποθέσεων και ιδρυμάτων. Άρα υπάρχει τέτοια σύγκρουση αρμοδιοτήτων και στην τελική ανάλυση κάπου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφασίζεται ποιο θα είναι αρμόδιος και δεν θεωρώ ότι είναι πάντα σαφέ το πώ λαμβάνονται οι φάσεις αυτέ. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν χρονικέ προθεσμίε, ή άλλω τραβούν προβολικά σε μάκρο οι εκθέσει πρωτοβουλία. Μάλιστα. Άρα το άρθρο 51 θεωρώ ότι έχει σκοπό να επιλύσει ακριβώς τέτοιες διαμάχες οι οποίες μπορεί χωρίς να επιληθούν να συνεχίζονται για πάντα. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία γρήγορα μεταξύ των επιτροπών για την κατανομή των αρμοδιοτήτων αυτών δάλος Θα μας επιβάλλει μια λύση η διάσκεψη των Προέδρων. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορούμε να το συζητήσουμε και να το σκεφτούμε φυσικά περαιτέρω. Μία πρόταση τροπολογία την οποία κατήρτισα για να διευκρινίσω τη διατύπωση και μπορούμε λοιπόν να θέσουμε την προθεσμία στις 15 Μαρτίου για την κατάθεση τροπολογιών. Συμφωνείτε? 15 Μαρτίου λοιπόν το βράδυ προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Από ό,τι φαίνεται ολοκληρώσαμε, εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Έφτασε και ο συνάδελφος Μπροκ βέβαια, αλλά θα μας μιλήσει αύριο για το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της τροποποίησης των συνθήκων. Ε, ε, ναι, ε, μην ανησυχείς, εγώ απλώς ήθελα να σε χαιρετήσω ιδιαίτερος. Αύριο θα μας μιλήσει και για το θέμα το πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν 9 η ώρα με τους συντονιστές. Μετά θα έχουμε την Αντιπρόεδρο Wallis που θα μας μιλήσει για το θέμα της διαφάνειας, το μητρό της διαφάνεια, διαφάνειας και μετά θα μας μιλήσουν οι συνάδελφοι Μπρόκ και Γκουελτιέρη γύρω στις 10 και μισή για την τροποποίηση των συνθήκων. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα τα ξαναπούμε.